Αγαπητοί συνάδελφοι, προτείνω να ξεκινήσουμε τις εργασίες μας. Σας θυμίζω ότι αυτό το σεμινάριο επικεντρώνεται απόλυτα στα προβλήματα της συμπληρωματικότητας ανάμεσα στους εθνικούς προϋπολογισμούς και στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό και όλος ιδιαίτερος στο ρόλο των διαθροτικών ταμείων και του Ταμείου Συνοχής στο πλαίσιο της υλοποίησης των στόχων του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου σε επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έπειτα σε επίπεδο του κάθε κράτους μέλους, όσον αφορά δηλαδή τους εθνικούς στόχους. Θα ήθελα να χαιρετήσω ε, τον πρόεδρο Φίλιππο Σαχινίδη, που είναι αντιπρόεδρος της Επιτροπής ε, Οικονομίας και ε, απολογισμού και γενικού ισολογισμού του κράτους και ελέγχου της εκτέλεσης του προπολογισμού του κράτους της Ελλάδας και που είναι ε, συμπρόεδρος της σημερινής συνεδρίασης ε, με εμένα, τον Αλέν Λαμασούρ, που, είμαι πρόεδρος της Επιτροπής Προϋπολογισμού του Ευρωκοινοβουλίου. Να μιλήσω και να παρουσιάσω την κυρία Μαρία Ντελμάρ Αγκούλο Μαρτίνες, γερουσιαστή της Επιτροπής Οικονομίας και Δημόσιας Δίκησης του Γερουσίας της Ισπανίας, ε, τον κύριο ε, κύριε Μπιρούτ Μπερβερσάιτε, μέλος της Επιτροπής Οικονομίας και της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων του ΣΕΙΜΑΣ της ε, Βουλής της Δημοκρατίας της Λιθουανίας. Και μετά τον κύριο Βάλτερ Ντεφά, που είναι Γενικός Διευθυντής υπεύθυνο για την ε, περιφερειακή και αστική πολιτική της, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Να θυμίσω πως όλοι όσοι είναι παρόντες και επιθυμούν να πάρουν το λόγο, να θέσουν ερωτήσεις ή να κάνουν παρατηρήσεις μετά από τις εισηγήσεις καθενός από τους προσκεκλημένους μας, θα πρέπει να συμπληρώσει το έντυπο που σας έχει διανεμηθεί, ούτω ώστε να μπορέσουμε να δώσουμε το λόγο σε όλους όσους το επιθυμούν και ο κανόνας επί το οποίο έχουμε συμφωνήσει και που ίσχυσε εχθές για τις Ολομέλειες αλλά και θα ισχύσει και σήμερα για κάθε ένα από τα εργαστήρια είναι δύο εθνικοί βουλευτές, ένας ευρωβουλευτής. Και θα προσπαθήσουμε βεβαίως με τον συμπρόεδρο σεχενίδη να εξασφαλίσουμε την πολιτική και γεωγραφική ισορροπία εάν τεθεί τέτοιο πρόβλημα. Δύο λόγια εισαγωγικά από μέρους μου. Αυτή η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα διοργανώνεται μέσα στο πλαίσιο της διαδικασίας που αποκαλείται Ευρωπαϊκό Εξάμεινο και για τα εμπλεκόμενα κράτη-μέλη στο πλαίσιο της εφαρμογής της Συνθήκης Δημοσιονομικής Σταθερότητας που προβλέπει την ε, σύγκληση διακοινοβουλευτικών συνεδριάσεων, διασκέψεων, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί ο κοινοβουλευτικός έλεγχος, η δημοκρατική παρακολούθηση και η δημόσια συζήτηση για τις θέσεις που λαμβάνονται είτε υπό τον τίτλο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης των 28 κρατών μελών, είτε υπό την συνθήκη σταθερότητας ε, για τα κράτη μέλη που ε, εμπλέκονται, που διέπονται μάλλον από αυτήν. Εμείς συμφωνήσαμε με την Ελληνική Προεδρία, ούτω ώστε μετά τις ολομέλειες που έγιναν τη Δευτέρα και χτες, σήμερα το πρωί να εργαστούμε ε, σε εργαστήρια, σε σεμινάρια ε, που αντιστοιχούν σε τρεις διαφορετικές ε, ανησυχίες διαστάσεις μάλλον αυτού του θέματος. Το πρόβλημα του συντονισμού των οικονομικών πολιτικών στην Νομισματική Ένωση, το πρόβλημα της ε, κοινωνικής πολιτικής, με κοινωνική διάσταση δηλαδή, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και εδώ το θέμα της συμπληρωματικότητας ή παραπληρωματικότητας των προϋπολογισμών ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός στην ουσία είναι ο 29ος προϋπολογισμός της Ένωσης. Πρόκειται για έναν μικρό προϋπολογισμό όσον αφορά το καθάριστο εγχώριο προϊόν. Είναι το 1% του ακαθόριστου εγχωρίου προϊόντος της Ένωσης, αλλά πρόκειται για ένα σημαντικό προϋπολογισμό όσον αφορά τον οικονομικό του αντίκτυπο, διότι το 94% του προϋπολογισμού της Ένωσης το οποίο η τάξη μεγέθους είναι 140 δις. Το 94% λοιπόν της 100 εξ αυτών είναι αφιερωμένα σε οικονομικές επεμβάσεις και επενδύσεις Άρα λοιπόν είναι μια μεγάλη διαφορά με τους εθνικούς μας ε, προϋπολογισμούς όπου οι λειτουργικές δαπάνες τους είναι πολύ πιο ψηλές για ιστορικούς λόγους και γιατί υπάρχουν μεγάλες δημόσιες υπηρεσίες πολύ δαπανηρές όπως είναι η παιδεία, η άμυνα, η κοινωνική πρόνοια και αυτά εμπίπτουν στις εθνικές αρμοδιότητες και όχι στις κοινοτικές. Αυτό σημαίνει ότι σε μια περίοδο όπως αυτή που διανύουμε, όπου το σύνολο της Ένωσης βρίσκεται στα πρόθυρα της ύφεσης και ταλαντεύεται ανάμεσα στην ύφεση και την ανάκαμψη, πολλές χώρες, ε, μεταξύ των οποίων δυστυχώς η Ελλάδα διανύουν ε, σοβαρή ύφεση εδώ και πολλά χρόνια και το, ο μέσος όρος της Ένωσης ε, επίσης ταλαντεύεται, σε μια φάση όπου οι χώρες πρέπει να συνεχίσουν τις προσπάθειες σημαντικές που κάνουν για να βάλουν τάξη στη δημόσια οικονομία τους, ε, σε μια φάση όπου ε, επίσης πρέπει να κάνουν όλα τα κράτη τεράστιες προσπάθειες ανταγωνιστικότητας, οφείλουμε να προσπαθήσουμε να χρησιμοποιήσουμε καλύτερα αυτόν τον ευρωπαϊκό προπολογισμό που είναι προπολογισμό παρέμβαση και επενδύσεων για να συνοδεύσει τους εθνικούς προπολογισμού, ώστε να εξασφαλίσουμε εν ότι θα επιτευχθούν οι γενικοί στόχοι της Ένωσης. Διαθέτουμε λοιπόν ε, τον απολογισμό της εφαρμογής ε, ε, της υλοποίησης, των, της εκτέλεσης μάλλον των ταμείων, των διαρθρωτικών αλλά και του κοινωνικού ταμείου που είναι τα βασικά μέσα για να βοηθηθούν τα κρατημέλη, αντιπροσωπεύουν το 1 τρίτο με το 40% του προϋπολογισμού. Έχουμε λοιπόν αυτόν τον απολογισμό, τον ισολογισμό του για την περίοδο 2007-2013, που ήταν εξαιρετικά δύσκολη, ε, που χαρακτηρίστηκε από την κρίση. Και είναι πολύ ενδιαφέρον να παρατηρήσουμε τον τρόπο με τον οποίο αυτές οι πολιτικές μπόρεσαν να στηρίξουν την οικονομική δραστηριότητα, να διαπιστώσουμε ότι οι δυνατότητες χρήσης, απορρόφησης των πιστώσεων ήταν πολύ σημαντικέ σε ορισμένες χώρες, μικρότερες σε άλλες, ότι ε, για να μπορέσουμε να προσαρμο... όταν μάλλον για να μπορέσουμε να προσαρμοστούμε στην εξέλιξη της κρίσης θελήσαμε να επαναπροσανατολίσουμε τα... τις πιστώσεις προς άλλα προγράμματα με πιο άμεσο αντίκτυπο ή με πιο μακροπρόθεσμο αντίκτυπο στην ανταγωνιστικότητα όπως είχε προτείνει ο πρόεδρος Βαρόζο. Αυτό πέτυχε σε κάποιες χώρες αλλά λιγότερο καλά πήγε σε άλλες. Και γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό να έχουμε την μαρτυρία, τις μαρτυρίες όλων. Τι πήγε καλά, τι δεν πήγε καλά, ε, ήταν καλό το σύστημα που φτιάξαμε ή όχι. Και έπειτα πέρυσι Διαπραγματευτήκαμε και εμείς εδώ στο Ευρωκοινοβούλιο με την Επιτροπή ε, ε, Περιφερειακών ε, Υποθέσεων ήμασταν στην πρώτη γραμμή. Φτιάξαμε το νέο πρόγραμμα για το 2014-2020. Φέτος είναι η πρώτη χρονιά αυτού του προγράμματος. Πήγε καλά. Πώς προετοιμάζονται τα νέα εθνικά προγράμματα στις διάφορες χώρες με βάση αυτό το νέο πλαίσιο σε πολλές, μάλλον ανάμεσα στις προτάσεις που έχουμε κάνει Ο αριθμός των προγραμμάτων και η κατανομή των κονδυλίων ανάμεσά τους σε ποιότητα και ποσότητα είναι η ίδια σε όλες τις χώρες, είναι ικανοποιητική, γιατί σε κάποιες χώρες υπάρχει μέγας κατακαιρματισμός. Και αν διαχέονται τα κονδύλια σε δεκάδες χιλιάδες προγράμματα, ο αντίκτυπος οικονομικός είναι ο ίδιος, όπως αν τα συγκεντρώναμε σε μια, καμιά δεκαριά μεγάλα προγράμματα. Θα ήταν ενδιαφέρον να ακούσουμε το σύνολο λοιπόν των εμπειριών και των μαρτυριών σας ε, που ε, ποικίλουν ανάλογα με τη χώρα και φυσικά και η ποιότητα του προγράμματος ε, παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Αυτά λοιπόν είναι τα προβλήματα που, τα ερωτήματα που τίθενται και καταρχήν θα δώσω το λόγο στους ε, ομιλητές μας που έχουν 5 με 10 λεπτά έκαστος για να παρουσιάσουν την άποψη της χώρας τους ή στο πλαίσιο της Επιτροπής του ε, οργανισμού που αντιπροσωπεύουν και μετά θα γίνει η συζήτηση με τους βρισκόμενους στην αίθουσα. Θα δώσω λοιπόν το λόγο καταρχήν στον κύριο Ντέφα, που είναι γενικό Διευθυντής της Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε και κύριοι. Είμαι ιδιαίτερα ευγνώμων για την πρόσκληση στην πολύ σημαντική αυτή συνεδρίαση των ε, Εθνικών Βουλευτών με τους Ευρωβουλευτές. Επ' ευκαιρία θα ήθελα να ευχαριστήσω και την Επιτροπή Προϋπολογισμών για την υποστήριξή της ε, στην πολιτική συνοχή. Γιατί χάρη σε αυτήν ε, μπορέσαμε πέρυσι να χρησιμοποιήσουμε ένα προϋπολογισμό των 43 δισεκατομμυρίων που είναι ιστορική σημασία προϋπολογισμός για τις περιφέρειες και μάλιστα μας περίσσεψαν 19 δισεκατομμύρια που δεν είχαμε πληρώσει στο τέλος του χρόνου γιατί δεν είχαμε αρκετές πιστώσεις. Οπότε θα χρειαστούμε περαιτέρω υποστήριξη από την Επιτροπή σας και στο μέλλον. Και περνάω στα αγγλικά. Σήμερα θα μιλήσω για τον ρόλο που διαδραματίζουν τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία, τα ESI όπως λέμε, για το ρόλο που διαδραμάτισαν στο παρελθόν και που θα συνεχίσουν να παίζουν για να στηρίξουν την ανάπτυξη και τη θέση απασχόληση σε ένα ριζικά διαφορετικό οικονομικό περιβάλλον. Οι αλλαγές αυτές οι ρηξικέλευτες στο οικονομικό περιβάλλον οφείλονται στη βαθύτατη οικονομική κρίση που ήταν άνευ προηγουμένου για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και μάλιστα πρόκειται για ένα μεταβαλλόμενο περιβάλλον, καθώς ε, μετά την κρίση έχει αλλάξει ο τρόπος χάραξη των πολιτικών, των οικονομικών πολιτικών. Σήμερα έχουμε έναν πολύ καλύτερο συντονισμό οικονομικών πολιτικών σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όπως περιχαρακώνεται από το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο. Εγώ λοιπόν θα κάνω μια σύντομη ανακεφαλαίωση των μέχρι τώρα ενεργειών μας προκειμένου να ενισχύσουμε την ανάπτυξη και την απασχόληση για την περίοδο 2007-2013 που ήταν η προηγούμενη περίοδος προγραμματισμού και στο δεύτερο τμήμα της ε, ομιλίας μου θα σας ε, περιγράψω την οργάνωσή μας για τη νέα περίοδο 2014-2020. Μπορούμε να περάσουμε παρακαλώ στην επόμενη διαφάνεια. Ευχαριστώ. Στο παρελθόν και με την κρίση, τα διάφορα οικονομικά μοντέλα που είχαμε έδειξαν ότι η πολιτική συνοχής αύξησε το ΑΕΠ κατά 1% και παραπάνω κατά μέσο όρο στις βασικές χώρες δικαιούχους. Θα μπορούσε κανείς να πει, «Εχει και τι είναι 1% ελάχιστο, αλλά 1% του ΑΕΠ δεν είναι αμεληταίο ποσοστό. Ιδιαίτερα όταν λάβει κανείς υπόψη το γεγονός ότι η συνολική συμβολή στην Επιτροπή Συνοχής είναι μόνο 0,3% του συνολικού κοινοτικού ΑΕΠ. Οπότε, στις βασικές χώρες αποδέκτες, το ΑΕΠ θα ήταν πάνω από 1% χαμηλότερο, χωρίς τις ενέργειες, τις παρεμβάσεις της πολιτικής συνοχής. Για να είμαστε όμως λίγο πιο συγκεκριμένοι, ε, σας παρουσιάζω εδώ μερικά βασικά επιτεύγματα της περίοδου 2007-2012. Αυτά είναι τα πιο πρόσφατα στοιχεία που έχουμε και είναι αρκετά εντυπωσιακά Βλέπετε πόσες χιλιάδες θέσεις απασχόλησης δημιουργήθηκαν, πόσες ε, εταιρείε στηρίξαμε, ε, σιδηροδρομικές γραμμές, πόσοι αυτοκινητόδρομοι κατασκευάστηκαν, ε, μεγαλύτερη πρόσβαση στο ευρυζωνικό διαδίκτυο, πρόσβαση πολιτών σε καθαρό πόσιμο είδωρ. Πολύ σημαντικό. Και μάλιστα το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο αριθμίσε 15 εκατομμύρια μέλη και ανθρώπους που συμμετείχαν στις δράσεις τους κάθε χρόνο. Είναι πολύ σημαντικό και εντυπωσιακό νομίζω αυτό το ποσό. 15 εκατομμύρια άνθρωποι το χρόνο συμμετείχαν σε δράσεις του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Η πολιτική συνοχή ε, μάλιστα στήριξε την ανάπτυξη και τις θέσεις απασχόλησης ακόμη και στην περίοδο της κρίσης. Αυτό που όμως είναι ατυχές και δημιουργεί τεράστια πρόκληση είναι ότι οι ανισότητε μεταξύ των πλέον ανεπτυγμένων περιοχών και των λιγότερων ανεπτυγμένων περιφερειών έχει αυξηθεί για πρώτη φορά. Πριν την κρίση είχαμε μια θετική τάση με μείωση των ανισοτήτων μεταξύ των ε, πιο ανεπτυγμένων και των λιγότερο ανεπτυγμένων περιφερειών. Τώρα δυστυχώς με την κρίση έχουν ε, ενισχυθεί αυτές οι ανισότητες, κάτι που δημιουργεί πρόκληση στην πολιτική συνοχή. Ποιες ήταν όμως οι συγκεκριμένες μας ε, αντιδράσεις στην κρίση. Τα προγράμματα για την περίοδο 2007-2013 είχαν χαραχθεί και προγραμματιστεί πριν από την κρίση. Είναι σαφές λοιπόν ότι με την κρίση δημιουργήθηκε μια ρηξικέλευτη αλλαγή στην κατάσταση και φυσικά κληθήκαμε να προσαρμοστούμε σε αυτές τις μεταβολές. Η πολιτική συνοχής λειτουργεί με τέτοιο τρόπο ώστε τα κοινοτικά κονδύλια συγχρηματοδοτούν κάποιες ε, εθνικές δαπάνες. Πρόκειται για το σύστημα της ε, κοινή διαχείρισης. Με την κρίση όμως, οι τοπικοί, περιφερειακοί και εθνικοί προϋπολογισμοί υπέστησαν τεράστιες ε, πιέσεις για εξυγίαση, οπότε χρειάστηκε και εμείς να αντιδράσουμε και το κάναμε αυξάνοντας το ποσοστό κοινοτικής συγχρηματοδότησης, ώστε να διευκολύνουμε και να ανακουφίσουμε κάπως τους εθνικούς προϋπολογισμούς. Αυξήσαμε λοιπόν και τις προκαταβολές το 2009 ε, με 6,2 δισεκατομμύρια επιπλέον. Αυξήσαμε στο μέτρο του δυνατού τη συγχρηματοδότηση, το ποσοστό της συγχρηματοδότησης ε, προσθέτοντας 29 περίπου δισεκατομμύρια και για τις ε, χώρες προγραμματισμού αυξήσαμε ακόμη και το μέγιστο ποσοστό συγχρηματοδότησης ε, στο 95%, κάτι που έφερε ακόμη 1,8 σχεδόν 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Οπότε ανταποκριθήκαμε στην δυσχερή οικονομική κατάσταση και δημοσιονομική κατάσταση των κρατών μελών. Και με την συρρήκνωση της οικονομικής δραστηριότητας ε, κρίση δεν είχε πια νόημα να προωθήσουμε μόνο τις επιχειρήσεις, να στηρίξουμε μόνο τις επιχειρήσεις και την καινοτομία ε, σε προϊόντα και τρόπους παραγωγής. Έπρεπε να βοηθήσουμε και απλές ε, επιχειρήσεις, γιατί αυτές ήταν που βρέθηκα σε πολύ δύσκολη θέση εξαιτία έλλειψης πρόσβασης ε, προς τη χρηματοδότηση. Κόπηκε ο δρόμος προς τη χρηματοδότηση. Γι' αυτό και τροποποιήσαμε τον κανονισμό προκειμένου να διαβρύνουμε το πεδίο εφαρμογή τη επιλεξιμότητα για το εργασιακό κεφάλαιο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, για παράδειγμα, που έγιναν επιλέξιμε, ενισχύθηκαν τα χρηματοοικονομικά εργαλεία για να, περιλαμβάνει και ε- περιλαμβάνουν και την ενεργειακή αποδοτικότητα, την κοινωνική στέγη και ούτω καθεξής. Διευρύνθηκε λοιπόν η επιλεξιμότητα για να προσαρμοστούμε καλύτερα στην κρίση. Και όπως είπε ο πρόεδρος της Επιτροπής Προϋπολογισμών, έπρεπε να προσαρμόσουμε τα προγράμματα και να κατευθύνουμε τα κονδύλια εκεί που χρειάζονται περισσότερο. Έγινε ένας αναπρογραμματισμός της τάξης των 45 δισεκατομμυρίων ευρώ, δηλαδή περίπου 13% των προγραμμάτων. Και όπως θα θυμάστε, είχαμε κάποιες δράσεις για την ανεργία των νέων και την υποστήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε 8 χώρες μέλη το 2012 και όλες αυτές οι δράσεις βοήθησαν περίπου ένα εκατομμύριο νέους και 50.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Βλέπετε λοιπόν ότι η πολιτική συνοχής έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο προκειμένου να ανταποκριθεί στις ανάγκες που δημιούργησε η κρίση και να συνέχισε να στηρίζει και να προωθεί την ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Οφείλω πάντως να ομολογήσω ότι όλα αυτά έγιναν κάπως γρήγορα, σαν να προσπαθούσαμε να, βι... να σβήσουμε μια φωτιά, ένα πυροσβεστικό και άμεσο τρόπο, αλλά είναι φυσιολογικό όταν έχει, κανείς όταν έχει κάποιος να αντιμετωπίσει μια κρίση και μια αναπάντηχη κατάσταση. Τώρα, στην επόμενη περίοδο προγραμματισμού, η πολιτική συνοχής, κατά τη γνώμη μας, θα αποτελέσει σημαντικό πυλώνα των οικονομικών πολιτικών και θα ήθελα να σας ε, περιγράψω το μείγμα πολιτικών ε, στο Ευρωπαϊκό Εξάμεινο χρησιμοποιώντας ε, το σχήμα του τριγώνου. Έχουμε λοιπόν στην κορυφή την δημοσιονομική εξυγίαση, γιατί χωρίς υγιή δημόσια οικονομικά δεν νοείται υγιής οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη. Έχουμε στη μία γωνία του τριγώνου την ανάγκη διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων. Σε πολλές χώρες με η λειτουργία της ε, αγοράς, ακόμα και της αγοράς εργασίας θα πρέπει να βελτιωθεί, να βελτιωθούν τα εκπαιδευτικά συστήματα, η καινοτομία, τα συστήματα καινοτομίας και έρευνας, προκειμένου να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και της οικονομίας. Επίσης τα κοινωνικά συστήματα έπρεπε να προσφέρουν προσαρμοστούν στις δημογραφικές αλλαγές. Βέβαια, η δημοσιονομική εξυγίαση και οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις δεν αρκούν από μόνα τους. Γιατί έτσι δεν έχουμε τρίγωνο. Είναι σαν να έχουμε μια καρέκλα με δύο μόνο πόδια για να στηριχθεί, να έχει ισορροπία η καρέκλα, χρειάζεται και τρίτο πόδι και αυτή είναι η άλλη γωνία του τριγώνου που είναι η στήριξη της ανάπτυξης και της ε, επένδυσης. Και εκεί βρίσκουμε το ρόλο των Ευρωπαϊκών Διορθωτικών και Επενδυτικών Ταμείων. Στο μέλλον, λοιπόν, ο ρόλο των Ευρωπαϊκών Διορθωτικών και Επενδυτικών Ταμείων θα αποτελέσει ένα απόσπαστο τμήμα του μείγματο πολιτικών. Βέβαια, το ένα τρίγωνο δεν απαρτίζεται μόνο από τρει γωνίε. Χρειάζεται και πλευρέ που να ενώνουν αυτέ τι γωνίε. Και αυτέ οι πλευρέ, αυτέ οι γραμμέ που ενώνουν τι γωνίε, δείχνουν του δεσμού μεταξύ των διαφόρων σημείων κορυφών του τριγώνου. Και είναι κάποια στοιχεία της επόμενης προγραμματικής περίοδου. Για παράδειγμα, βλέπουμε το σύνδεσμο μεταξύ δημοσιονομικής εξυγίασης και παρότρησης ανάπτυξης και επένδυσης. Έχουμε την περίφημη μακροοικονομική αιρεσιμότητα. Αν μια χώρα επανειλημμένως δεν τηρήσει τις υποσχέσεις που έχει λάβει στα πλαίσια της διαρθρωτικής εξυγίασης, δεν μπορεί να το κάνει χωρίς να υφίσταται τις συνέπειες ε, από τη χρηματοδότηση των ταμείων. Επίσης, ελπίζουμε ότι με την ε, δημοσιονομική εξυγίανση δαπάνες ε, που είναι φιλικές προς την ανάπτυξη και την απασχόληση θα διασφαλιστούν. Επίσης υπάρχει ένας σύνδεσμος μεταξύ της πλευράς ανάπτυξης και επένδυσης και ανάπτυξης και των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων. Και εκεί έχουμε την ε, εξάντε Και χρειαζόμαστε κάποιους όρους και προϋποθέσεις που θα πρέπει να συντρέχουν. Τότε και μόνο τότε έχει νόημα η επένδυση σε συγκεκριμένα προγράμματα, γιατί τότε μόνο θα είναι αποδοτικές οι επενδύσεις. Για παράδειγμα, πριν ε, χρηματοδοτήσουμε κάποιους ε, σταθμού αποτέφρωσης, για παράδειγμα αποβλήτων, θα πρέπει να είμαστε βέβαιοι ότι υπάρχουν κάποια στοιχεία, ε, προγράμματα διαχείριση των αποβλήτων. Για παράδειγμα, αν θα γίνεται ανακύκλωση των αποβλήτων. Όταν θέλουμε να στηρίξουμε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, έχει αυτό νόημα σε ένα επιχειρησιακό περιβάλλον που είναι φιλικό Προ τι ε, επιχειρήσει. Δεν έχει νόημα να στηρίζουμε επιχειρήσει σε ένα εχθρικό επιχειρησιακό περιβάλλον, επιχειρηματικό περιβάλλον. Οπότε γίνεται μια τέτοια εκ των προτέρων αιρεσιμότητα. Και μόνο εφόσον συντρέχουν οι προποθέσει αρχίζει η ροή των κεφαλαίων. Βέβαια και στην τρίτη πλευρά έχουμε ένα σύνδεσμο, γιατί τα διαρθρωτικά ταμεία στηρίζουν τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις με τεχνογνωσία, με, για την ανάπτυξη ανάπτυξη στρατηγικών μεταφορών ή διαχείριση των αποβλήτων, για παράδειγμα. Οπότε έτσι οι πλευρές του τριγώνου κρατάνε τις κορυφές μαζί και έτσι έχουμε το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο με τις ειδικές συστάσεις αναχώρα. Αν λοιπόν θέλουμε η πολιτική συνοχή να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο για την ανάπτυξη και την απασχόληση, θα πρέπει να προσανατολίζεται προς τα αποτελέσματα. Και περνάμε στην επόμενη διαφάνεια. Η πολιτική μας θα πρέπει να στοχεύει σε αποτελέσματα. Τι σημαίνει αυτό για την ανάπτυξη και την απασχόληση. Σημαίνει συγκέντρωση. Το είπαν οι Γερμανοί. Θεματική συγκέντρωση, και οικονομική συγκέντρωση σε κινητήριους μοχλούς της ανάπτυξης, δηλαδή στην έρευνα, καινοτομία, τεχνολογική ανάπτυξη, μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ε, οικονομίες χαμηλής χρήσης άνθρακα, αγορά εργασίας, ε, κοινωνική ένταξη, ανθρώπινο κεφάλαιο. Θα έλεγε κανείς ότι αυτή είναι, παρά είναι γενική προσανατολισμή. Και έχει δίκιο. Παρ' όλα αυτά θα πρέπει να είναι πηγή έμπνευση για τα μεμονωμένα προγράμματα που αυτά θα είναι εξατομικευμένα, θα είναι προσαρμοσμένα στις ανάγκες. Και έτσι επαναρχόμαστε στο Ευρωπαϊκό Εξάμεινο. Τα προγράμματα για συγκεκριμένη χώρα θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαιτερότητες της χώρας και τις ειδικές συστάσεις της χώρας αυτής. Επίσης θα πρέπει να είναι προσαρμοσμένα τα προγράμματα στις τοπικές και εθνικές ανάγκες. Και γι' αυτό έχουμε στρατηγικές έξυπνης εξειδίκευσης. Εκεί έχουμε σημαντική συμμετοχή των τοπικών κοινοτήτων, πανεπιστημίων, επιχειρηματιών και ούτω καθεξής. Θα πρέπει λοιπόν τα προγράμματα να περιέχουν σαφή ορισμό για τα αποτελέσματα που θέλουν να πετύχουν. Θέλουμε ε, σημαντικούς ε, ρωμαλαίους δείκτες για να μπορούμε να ελέγχουμε και να παρακολουθούμε τα προγράμματα, να κάνουμε την αξιολόγηση και με το πλαίσιο για την απόδοση και το αποθεματικό απόδοσης θα κατευθύνουμε τα κονδύλια μας ε, προκειμένου να γίνεται καλύτερη χρήση του, να πιάνουν τόπο και να έχουν και την καλύτερη έκβαση. Και με την εκ των προτέρων αιρεσιμότητα θα έχουμε πια και τις προϋποθέσεις για αποτελεσματικές επενδύσεις. Φέτος, ε, το 2014, θα έχουμε μια χρονιά ορόσημο για τη διαδικασία αυτή. Γιατί φέτος, το 2014, θα γίνει η υποβολή και η έγκριση των προγραμμάτων. Και αυτά τα προγράμματα θα διαμορφώσουν το πλαίσιο για την ε, τόνωση της ανάπτυξης και, την και της απασχόλησης. Πέρυσι είχαμε την υιοθέτηση της νομοθεσίας. Έχουμε πλέον 325 δισεκατομμύρια για την πολιτική συνοχή για το 2014-2020 και το, έχουμε το Ταμείο Γεωργικής Ανάπτυξης και μαζί με το Ταμείο Αλία ξεπερνάμε τα 400 δισεκατομμύρια, αν προσθέσουμε και αυτά τα δύο ταμεία. Βλέπετε ότι είναι πολύ σημαντικό αυτό το ποσό. Οπότε στο πρώτο στάδιο τα, κράτη-μέλη θα υποβάλουν τις συμφωνίες εταιρική σχέσης, το γενικό έγγραφο στρατηγικής τους δηλαδή, και εκεί θα πρέπει να δείξουν πώς θα λάβουν υπόψη τις ειδικέ συστάσεις ανά χώρα. Και κάτι άλλο πολύ σημαντικό είναι ότι αυτές οι αναπτυξιακές πολιτικές και αυτές οι συμφωνίες εταιρική σχέση θα πρέπει να στηρίζονται σε μια ευρύτερη εταιρική σχέση ενδιαφερομένων στα κράτη-μέλη. Και όσο προχωρεί το έτος, θα έχουμε και τα επιχειρησιακά προγράμματα, τα λειτουργικά προγράμματα που θα υποβληθούν και θα εγκριθούν και θα είναι τα έγγραφα προγραμματισμού για να συγκεκριμενοποιηθούν οι στόχοι και για να έχουμε χρηστή δημοσιονομική διαχείριση και να επιτύχουμε την ανάπτυξη και την απασχόληση. Όλοι πια είμαστε ενωμένοι και συνεργαζόμαστε για μια, σε μια κοινή προσπάθεια σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και κοινοτικό επίπεδο προκειμένου να βάλουμε σε σωστές γραμμές αυτά τα προγράμματα και να έχουμε τη μέγιστη απόδοσή τους ώστε να έχουμε έξυπνη, βιώσιμη, αηφόρο και ανάπτυξη που δεν θα αποκλείει κανέναν. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε όπως στο παρελθόν, σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Θα πρέπει να, να δώσουμε νέους προσανατολισμούς, σωστούς προσανατολισμούς και γι' αυτό ζητώ και τη δική σας υποστήριξη σε αυτήν την κοινή προσπάθεια. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Γενική Διευθυντά για την σαφίστατη σας εισήγηση. Ο κύριος Αχινίδης. Thank you very much. Representing the Hellenic Parliament. Εκπροσώπω το Ελληνικό Κοινοβούλιο και καλωσορίζω όλους ε, τους ε, συμμετέχοντες από τα εθνικά και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο γιατί θεωρώ ότι όλες οι συναντήσεις που λαμβάνουν χώρα εντός αυτής της ε, διακοινοβουλευτικής εβδομάδας είναι πολύ ουσιώδη, όχι μόνο για στενή επαφή μεταξύ εθνικών και ευρωβουλευτών, αλλά για περαιτέρω βελτίωση της ε, ε, αχθήσης διαδικασίας του Ευρωπαϊκού Εξαμενού. Πιστεύω ότι όλοι συμφωνούμε ότι αυτή η αλληλεπίδραση μεταξύ μας συμβάλλει στην καλύτερη αλληλοκατανόηση της δουλειάς του καθενός και θα μπορούσε να ευνοήσει τις προσπάθειές μας για καλύτερη προσπάθεια συντονισμού των οικονομικών πολιτικών στα πλαίσια αυτά. Το θέμα της συζήτησή μας είναι πολύ ενδιαφέρον, αναγκαίο και χρήσιμο. Η κρίση εστίασε την προσοχή της κοινή γνώμης την ε, προσπάθεια δημοσιονομικής εξυγίανσης, ε, τις περικοπές περιπολισμών και την ανάγκη για δύσκολες και κοινωνικά επίπονες διαφορετικές μεταρρυθμίσεις. Και επιπλέον, η έννοια του ενωσιακού προπολισμού κυρίως συνδέεται με σκληρές μάχες μεταξύ κρατών μελών και θεσμών, ε, με αντιπαραθέσεις μεταξύ αυτών που λαμβάνουν περισσότερα από όσα συμβάλλουν και ε, το, τον, αυτό που κάνουν το αντίστροφο. Μπορεί να έχει μικρές διαστάσεις, αλλά ο προπολογισμό και οι πολιτικές κλειδιά όπως οι διαστροτικές και οι δαπάνες συνοχής που είναι στο κέντρο της προσοχής μας ε, προσφέρουν πολύ προστιθέμενη αξία. Ιδιαίτερα η πολιτική συνοχής είναι το κύριο εργαλείο επενδύσεων για να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας, ανάπτυξη και κοινωνική συνοχή επίσης είναι σαφές, είναι μια πολιτική για αυτούς που την χρειάζονται περισσότερο. Η πολιτική συνοχής ήταν ο ακρογωνιαίος λίθος του σχεδίου Ευρωπαϊκής Ανάκαμψης που εγκρίθηκε το 2008 και τα πρόσφατα μέτρα, όπως αύξηση της χρηματοδότησης, οι συμπληρωματικές πληρωμές και η δυνατότητα αναπρογραμματισμού και ε, Κοινή αντιμετώπιση των κινδύνων ε, αποδεικνύουν πόσο τα διευθυντικά ταμεία και τα ταμεία συνοχή έχουν συμβάλει στις προσπάθειες ανάκαμψης. Τα μέτρα αυτά ήταν και είναι πολύ ουσιώδη βοήθεια, χείρα βοηθείας στις τεράστιες προσπάθειε που έχει κάνει και η χώρα μου και οι πολίτες της για να αντιμετωπίσουν τι επιπτώσει της οικονομικής κρίση που έχει μετατραπεί και σε κοινωνική κρίση. Η πολιτική συνοχή στην Ελλάδα θα επενδύσει κατά την ε, ε, τωρινή περίοδο προγραμματισμού πάνω από 20 δις. Αυτή τη στιγμή πάνω από 60% των διαφορετικών και ταμείων συνοχής δαπανώνται για να δημιουργήσουν ανάπτυξη και ε, θέσεις εργασίας, να αντιμετωπίσουν την κρίση και να απαλύνουν ένα τμήμα των αρνητικών της συνεπειών όλες αυτές. Οι επενδύσεις κάνουν τη διαφορά και για την οικονομία και τους πολίτες μας. Ένας μεγάλος αριθμός προγραμμάτων από μεγάλης κλίμακας ε, δημόσια έργα μέχρι μικρές τοπικές πρωτοβουλίες εκτελούνται για να βελτιώσουν την καθημερινή ζωή των πολιτών και όλα αυτά γίνονται σε ένα πολύ δύσκολο πλαίσιο δημοσιονομικής προσαρμογής και παρατεταμένης ύφεσης της ελληνικής οικονομίας. Τα τελευταία 6 χρόνια χάσαμε 25% του ΑΕΠ μας. Η ανεργία αυτή τη στιγμή είναι 27% και η ανεργία των νέων είναι 64%. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, η εφαρμογή, η εκτέλεση των διαφορετικών και των ταμείων συνοχής μέχρι τώρα έχουν δημιουργήσει μεταξύ 135 και 140.000 θέσεις εργασίας. Άρα ε, έχουν συμβάλει πάρα πολύ στη δημιουργία θέσεων εργασίας σε μια συγκυρία όπου είναι πρωτόγνωρα τα επίπεδα ανεργίας στην Ελλάδα. Αν συγκρίνουμε τα στοιχεία αυτά με τα στοιχεία για την ανεργία και την φτώχεια δεν είναι τόσο εντυπωσιακά, δηλαδή με τις ανάγκες για να αντιμετωπιστούν αυτά τα προβλήματα, αλλά οι πόροι αυτοί οπωσδήποτε παίζουν ζωτικό ρόλο για την αντιμετώπιση των αρνητικών επιπτώσεων. Από την αρχή της κρίσης η πολιτική συνοχή είναι ο κύριος πόρος για δημόσια μεδί στην Ελλάδα για περίπου το 65% του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων της Ελλάδας. Εξαιρετικές καταστάσεις ε, απαιτούν εξαιρετικά μέτρα. Και αυτό συνέβη με τα διαρθρωτικά και τα μία συνοχή στην Ελλάδα. Υπήρχε μεγάλη ανάγκη να προσαρμοστούν οι διαθέσιμοι πόροι στη σοβαρότητα της κατάστασης και να αυξήσουμε όλα τα δυνατά περιθώρια στο μέγιστο. Ευτυχώς αυτό συνέβη με πολύ συγκεκριμένα και πολύ διαφορετικά μέτρα. Η πρωτοβουλία για τους νέους, εγγύηση για τις μικρομεσαίες, αναπρογραμματισμός και αύξηση του ποσοστού συγχρηματοδότηση, του συντελεστή συγχρηματοδότηση με τη βοήθεια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και φυσικά την τεράστια και πολύ σημαντική στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Για την πρωτοβουλία για τους νέους, για παράδειγμα, για την ανεργία των νέων. Βοήθησε τους νέους άνεργους και του πτυχιούχους να αποκτήσουν μια πρώτη εργασιακή εμπειρία. Είχαμε ένα πρόγραμμα δράσης, τέσσερα δις, για να βοηθήσουμε την επιχειρηματικότητα και την ε, ε, ε, εργασία για τους νέους. Στην συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τον αναπρογραμματισμό για να στηρίξουμε περαιτέρω με ένα δις τις μικρομεσαίες. Οι μικρομεσαίες είχαν επίσης το ταμπιο εγγύσεων με αυτά το, οι διαρθρωτικοί πόροι βοηθούν ε, τις ελληνικές τράπεζες να χρηματοδοτήσουν μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Δόθηκαν περίπου 1,5 δις και ο συντελεστής ε, συγχρηματοδότησης που όπως υπόθηκε πήγε 85% και στην πραγματική πληρωμή 10% επίσης προβλέπεται. Και όλα αυτά είχαν επίπτωση 848 εκατομμύρια μέχρι στιγμής από όλα τα ταμεία. Και επίσης ε, η αναπροσαρμογή για, την, ε, για τους ομίλους για την κατασκευή αυτοκινητοδρόμων και αυτή βοήθησε και δημιούργησε θέσεις εργασίας όλα αυτά τα μέτρα μας επέτρεψαν να περάσουμε από το τελευταίο για ποσοστά απορρόφησης στους πρώτους πέντε. Έτσι δόθηκε πραγματική ρευστότητα στην πραγματική οικονομία και ε, διατήρησαν επιχειρήσεις εν ζωή και ορισμένους εργαζόμενους που αλλιώς θα ήταν στην ανεργία στην εργασία. Φυσικά πρέπει να κάνουμε πολλά ακόμη για να γίνει πραγματικά ανταγωνιστική η ελληνική οικονομία, να μπορεί να δημιουργεί βιώσιμη ενεργεία και θέσεις εργασίας, δηλαδή για να επιτύχει τους στόχους της Ευρώπης 2020 και τους στόχους λοιπόν του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Αλλά το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο μας ε, δημιουργεί, να, μας βοηθά να βρούμε απαντήσεις. Και μόνο αν υπάρχει συντονισμός και στόχευση των προσπαθειών των χωρών μπορεί να έχουν το επιθυμητό αποτέλεσμα για την ανάπτυξη. Για να έχουμε αυτή ε, την προσπάθεια συντονισμού, συμφώνησαν τα κράτη-μέλη να υπάρχει ο ετήσιο κύκλο ε, του συντονισμού των οικονομικών πολιτικών, το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο, όπου υπάρχει στρατηγική ευθυγράμμιση των πολιτικών συνοχή. Δυστυχώ, χώρε όπω η Ελλάδα δεν είναι τμήμα αυτού του διαλόγου και της αλληλεπίδρασης. Δυστυχώς οι χώρες ε, που έχουν ε, πρόγραμμα προσαρμογής ε, δεν λαμβάνουν τέτοιες συγκεκριμένες εθνικές συστάσεις. Ελπίζουμε πολύ σύντομα αυτή η πολύ ουσιώδης διαδικασία θα σταματήσει να θυσιάζεται για να έχουμε διαφάνεια και οικονομική λογοδοσία. Θέλουμε η πολιτική συνοχή να συνδέεται καλύτερα με την οικονομική διακυβέρνηση. Τα προγράμματα θα πρέπει να συνάδουν με τα εθνικά προγράμματα μεταρρυθμίσεων και να στηρίζουν τις προτεραιότητες μεταρρυθμίσεων που καθορίζουν οι ε, εθνικές προτάσεις, ε, οι προτάσεις για κάθε μια χώρα που κάνει το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε σαν να σημαίνει τίποτα. Επειδή υπάρχουν τόσοι δημοσιονομικοί περιορισμοί, πρέπει οπωσδήποτε να δαπανίσουμε κάθε ευρώ με τον πιο ευφύ δυνατό τρόπο για την περίοδο 2014-2020 έχουν εισαχθεί προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται για να γίνουν εκταμιεύσεις. Πρέπει δηλαδή τα προγράμματα και επενδύσεις να έχουν τα επιθυμητά αποτελέσματα. Στην περίοδο 2014-2020 οι πόροι αυτοί θα πρέπει επίση να εστιάζονται σε λιγότερε προτεραιότητε κλειδιά για να υπάρχει η αναγκαία κρίσιμη μάζα, ούτω ώστε να υπάρχει ισχυρή συμμετοχή στην ανάπτυξη και τι θέσει εργασία. Επειδή οι χώρε αντιμετωπίζουν διαφορετικέ προκλήσει, το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο και οι συστάσει του, που επιμένω πρέπει να περιλαμβάνουν και τι ε, χώρε προγράμματο, πρέπει να είναι προσαρμοσμένε στην κατάσταση και τι ανάγκε σε κάθε κράτο μέλο. Στην Ελλάδα διαπιστώνουμε τα πρώτα αδύναμα ακόμη δείγματα ε, ανάκαμψης που θα μπορούσαν να μας βοηθήσουν να βγούμε από τη σύραγγα. Πολλά και δύσκολα ακόμη πρέπει να κάνουμε. Αλλά αυτό που μπορώ να σας πω σίγουρα από την εμπειρία μου είναι ότι ο ενωσιακός προπολογισμό με, ε, πρωτοπόρο τον προπολογισμό συνοχή μα βοήθησε πάρα πολύ στι προσπάθειε να υπερβούμε την κρίση. Τα κράτη-μέλη, κάθε κράτο μέλο πρέπει να εργαστεί σκληρά. Να κάνει αυτό πρέπει να κάνει. Να μάθει από τα λάθη του παρελθόντο και να αξιοποιήσει βέλτιστα ε, του απαραίτητου διαθέσιμου πόρου. Αξιοποιώντα πλήρω την στρατηγική ε, ενίσχυση και συμβουλέ των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων. Παράλληλα, τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα θα πρέπει να αφήσουν αρκετή ευελιξία στα κράτη-μέλη για να αντιμετωπίσουν τι δικέ του συγκεκριμένε ανάγκε, να ψάξουν να βρουν ε, που υπάρχει δυναμικό ανάπτυξη και να αξιοποιήσουν αυτή τη στρατηγική βοήθεια αποφεύγοντα δογματικέ και στενά γραφειοκρατικέ προσεγγίσει. Περισσότερη και καλύτερη Ευρώπη είναι ο κοινό μα στόχο, η απάντηση στην κρίση η Ευρωπαϊκή, τα ευρωπαϊκά και, συγγνώμη, το Ευρωπαϊκό και τα Εθνικά Κοινοβούλια ε, ασκώντα τι αρμοδιότητε του και συνδυάζοντα τι προσπαθίε του για να αξιοποιήσουν καλύτερα τα εργαλεία μέσω του ευρωπαϊκού προπολογισμού, όπω τα διαθροτικά ταμεία και τα ταμεία συνοχή, μπορούν να στρώσουν το δρόμο για περισσότερα αποτελέσματα και για πολιτικέ που να εστιάζονται περισσότερο στα αποτελέσματα και τι ανάγκε των πολιτών. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε για αυτή την πολύ σαφή και εντυπωσιακή παρουσίαση του ελληνικού παραδείγματος από τις σημαντικές προσπάθειες που έχει καταβάλει το ελληνικό κράτος και ο ελληνικός λαός για την καλύτερη χρήση των ευρωπαϊκών κονδυλίων. Και τώρα να δώσω το λόγο στην κυρία Μαρία Δελμάρα Αγκούλο Μαρτίνες. Παρακαλώ, κυρία μου. Gracias, señor presidente. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και καλημέρα σε όλους σας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω πρώτα απ' όλα όλους σας για την ευκαιρία που μου δίνετε να σας παρουσιάσω τη γνώμη μου σε ένα τόσο σημαντικό θέμα της Ευρωπαϊκής Οικοδόμης που είναι η πολιτική συνοχή. Μίζον εργαλείο για τη σύγκληση, τις επενδύσεις, την ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Και είναι σημαντική αυτή η ευκαιρία σε μια πολύ κρίσιμη στιγμή για την, ε, για την έξοδο από την κρίση για να δείξουμε ότι με την όθηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και με την προσήλωση ευρωπαϊκές ιδέες μπορούμε να προωθήσουμε μια δίκαιη και εύρωστη ανάπτυξη αξιοποιώντα ευκαιρίε μα και το κοινωνικό μα μοντέλο. Με την έναρξη του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου 2014 έχουμε ένα νέο δημοσιονομικό ορίζοντα, αλλά έχουμε και σημαντική πύρα, Την πύρα από τα επιτεύγματα της πολιτικής συνοχής, από τα διαρθρωτικά ταμεία που συνέβαλαν στην ανάκαμψη, την οικονομική ανάκαμψη, την έξοδο από την κρίση, λαμβάνοντας από υπόψη τις ανάγκες και τις προτεραιότητες των επιμέρους χωρών και των επιμέρους περιφερειών της Ευρώπης. Είναι ήταν μια πολύ χρήσιμη εμπειρία και ένα πολύ σημαντικό μάθημα και για το μέλλον και ευκαιρία να αναλύσουμε όλη αυτή την κατάσταση. Η οικονομική κρίση σίγουρα ήταν η πιο ε, δρυμία και σοβαρή. Ήταν ε, πρόκληση πρώτης τάξης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα ολέθρια αποτελέσματα της στην οικονομία, στα δημόσια οικονομικά και ιδιαίτερα στην πραγματική οικονομία με την καταστροφή θέσεων απασχόλησης, όλα αυτά απέτυχαν μια άμεση δράση για να αναχαιτιστεί η κρίση. Και εδώ εντάσσεται η δράση της Ένωσης με την πρώτη ανακοίνωση Ευρωπαϊκής Επιτροπής τον Οκτώβριο του 2008. Έτσι εφαρμόζονται διαρθρώσεις στα διάφορα ταμεία γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, είχε επίγνωση της ανάγκης των κρατών μελών ε, να ανακουφιστούν στις προσπάθειες και στα δημόσια οικονομικά τους. Και μάλιστα ήταν πολύ θετική η απόκριση των κρατών μελών στις μεταρρυθμίσεις αυτές. Ήταν όλο και μεγαλύτερε οι ανάγκε χρηματοδότησης, χρειαζόταν λοιπόν μια ελαστικότητα στην επιλεξιμότητα των δαπανών και μια ε, διεύρυνση του πεδίου εφαρμογή προκειμένου να καλυφθούν και νέε πρωτοβουλίε και προγράμματα και φυσικά ε, χρειαζόταν και ένα ε, επαναπροσανατολισμό των δαπανών και των επενδύσεων. Πολλέ χώρε μέλη επωφελήθηκαν από τι μεταρρυθμίσει στα διαρθρωτικά ταμεία, από την νέα ελαστικότητα των διαρθρωτικών ταμείων, προκειμένου να κάνουμε αλλαγέ, είτε σε συγκεκριμένε περιφέρειε, είτε σε συγκεκριμένου τομεί που είχαν πληγεί από την οξύτατη κρίση. Γενικώ προσπαθήσαμε να αντιμετωπίσουμε συγκεκριμένες διαρθρωτικέ αδυναμίες και να ενισχύσουμε κάποιες πτυχές που ίσως δεν είχαν ληφθεί δεόντως υπόψη. Είμαι πεπισμένη ότι η απασχόληση είναι η καλύτερη κοινωνική πολιτική και μάλιστα συνιστά αδιαφυσβήτητη προτεραιότητα της κοινωνικής πολιτικής. Γι' αυτό και θα πρέπει να αποτίσουμε φόρο τιμής ε, σε όλε τις πρωτοβουλίε που εκμεταλλεύτηκαν το υπάρχον πλαίσιο για να δημιουργήσουν νέε ευκαιρίε. Όλες οι δράσεις ε, είχαν στόχο την τόνωση του επιχειρηματικού πνεύματος και ε, αντιμετώπιση των αναγκών χρηματοδότησης ιδιαίτερα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και φυσικά των αυτοαπασχολούμενων γιατί σε πολλές χώρες και στην Ισπανία απέδειξαν ότι μπορούν να δώσουν και αυτή τη συμβολή τους στην απασχόληση, να επιβιώσουν και ήταν σημαντικό να εξασφαλίσουμε απρόσκοπτη πρόσβασή τους στη χρηματοδότηση. Θα ήθελα εδώ να τονίσω τη μεγάλη σημασία που είχαν όχι μόνο στην Ισπανία, αλλά σίγουρα και στην Ισπανία, ε, η δήλωση των μελών του Συμβουλίου στις 30 Ιανουαρίου του 2012 επί της πρωτοβουλίας Μπαρόζο. Εκεί αναφερόταν ως προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης η ανάγκη ενίσχυσης της απασχόλησης και κυρίως της ε, απασχόλησης των νέων. Εκεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανέλαβε τη δέσμευση από κοινού με τα κράτη-μέλη να μην φυστεί προσπαθειών προκειμένου να αποκατασταθεί η απασχόληση των νέων και να αφιερώσει κονδύλια στην ε, ενίσχυση της ε, απασχόλησης των νέων και σε μέτρα και ενάψματα για τη χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Και μάλιστα στην Ισπανία καταβάλουμε τεράστιες προσπάθειες για να υλοποιήσουμε αυτή την πρωτοβουλία. Έχουμε μια ομάδα δράσης με εκπροσώπους Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ισπανικής Δημόσιας Διοίκησης προκειμένου να θεσπίσουμε μέτρα και δράσεις για να υλοποιήσουμε αυτή την πρωτοβουλία και έχουμε και μια ομάδα παρακολούθησης για την ανακατανομή των κονδυλίων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και του Ευρωπαϊκού Αναπτυξιακού Ταμείου. Επίσης κάνουμε έναν αναπρογραμματισμό και προσπαθούμε να καταπολεμήσουμε πιο αποτελεσματικά την ανεργία των νέων και να ενισχύσουμε, να ενισχύσουμε πολιτικές για να δημιουργήσουμε θέσεις απασχόλησης. Επίσης, αποκατάσταση της πρόσβασης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στη χρηματοδότηση είναι πολύ σημαντικό και η δράση της ΕΤΕ και της ΕΚΤ. Αλλά θα πρέπει να αξιοποιήσουμε τις ευκαιρίες που δίνονται με πρωτοβουλίες όπως το Τζέρεμι και το Τζέσικα στην Ισπανία αξιοποιούμε στο έπακρο τις πρωτοβουλίες αυτές. Αυτά τα χρηματοπιστωτικά μέσα που ε, δημιουργήθηκαν με τα ταμεία, τα διαρθρωτικά, είναι πολύ σημαντικά. Επίσης υπάρχει δυνατότητα συμπερίληψης ε, σημαντικών προγραμμάτων σε επιχειρηματικά προγράμματα, όπως είναι το Τεχνολογικό Ταμείο σε περιοφέρειες σύγκλησης. Επίσης μιλήσαμε για την ε, προσήλωση όλων μας στο στόχο της ανάκαμψης, ε, της δημοσιονομικής εξηγήσης και της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης. Είναι σημαντική αυτή η δέσμευση και η προσήλωση, αλλά χρειάζεται και αποφασιστική δράση, συνεπής και συνεκτική από όλα τα κράτη-μέλη. Και στην Ισπανία, πέραν της ε, σημαντικής δημοσιονομικής εξηγίασης, πέραν της εξηγίασης των δημόσιων λογαριασμών και του χρηματοπιστωτικού συστήματος, και πέραν της θέσπης σημαντικών μέτρων για καλύτερη λειτουργία της δημόσιας διοίκησης, εγκρίνουμε και εφαρμόζουμε μία δεύτερη γενιά μεταρρυθμίσεων που θα συμβάλλουν στην αποκατάσταση της, χρημα... της πίστης, την ενίσχυση της απασχόλησης και την ανάκαψη της οικονομίας. Προσπαθούμε να ενισχύσουμε τον παραγωγικό μας ιστό. Δεν θα πρέπει να ξεχνούμε ότι στην Ισπανία μεταξύ 2008 και 2011 χάθηκαν περίπου 3.800.000 θέσεις απασχόλησης και έκλεισαν περίπου μισό εκατομμύριο επιχειρηματικές πρωτοβουλίες. Σήμερα η πρωταρχική μας πρόκληση είναι να αναχαιτήσουμε αυτή την απώλεια θέσεων απασχόλησης. Σήμερα έχουμε 147.000 ε, ανέργους λιγότερους από πέρυσι. Αυτή είναι η βασική μας πρόκληση, αλλά άλλη σημαντική πρόκληση είναι η ανασυγκρότηση, η αποκατάσταση αυτού, αποκατάσταση του παραγωγικού ιστού. Οι μεταρρυθμίσεις αυτές που στοχεύουν σε αυτή την ανάκαμψη και την αποκατάσταση, αυτή η στρατηγική για την επιχειρηματικότητα των νέων και την απασχόληση των νέων που εγκρίθηκε το 2013, ο νόμος για την υποστήριξη των επιχειρηματιών και οι εγγυήσει για την ενότητα της αγοράς ε, αποτελούν πρωτοβουλίες ε, της Ισπανικής κυβέρνησης. Χρειάζεται λοιπόν αποφασιστική δράση εκ μέρους των κρατών μελών αλλά και εκ μέρους των κοινοτικών θεσμικών οργάνων γιατί η ανάκαμψη θα πρέπει να στηριχθεί σε καλά προσανατολισμένες πολιτικές από τα κράτη-μέλη αλλά και η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να θεσπίσει συγκεκριμένα μέτρα που θα έχουν πολλαπλαστικό αποτέλεσμα και θα δημιουργήσουν πολύ σημαντικές συνέργειες. Επιπλέον, ε, η ευρωπαϊκή οικοδόμηση θα είναι πιο στεναρή αν αποδείξει ότι μπορεί να αντιμετωπίσει συγκεκριμένα προβλήματα της ε, καθημερινότητας των πολιτών. Γι' αυτό θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό να χρησιμοποιηθούν κονδύλια σε πρωτοβουλίες ε, για την καταπολέμηση της ενέργειας των νέων ή για την ε, διευκόλυνση της πρόσβασης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε χρηματοδότηση. Ε, θα πρέπει να δίνουμε συγκεκριμένες λύσεις σε πολύ τα προβλήματα. Γι' αυτό και θεωρώ απαραίτητη την ευελιξία, την ελαστικότητα και τις δυνατότητες επαναπροσανατολισμού και προσαρμογής των κονδυλίων στις τρέχουσες ανάγκες. Τα διαρθρωτικά ταμεία έγιναν πιο ελαστικά και άρα πιο χρήσιμα, γιατί έτσι φτάνουν πιο γρήγορα τα κονδύλια και μάλιστα εξυπηρετούν καλύτερα τις ανάγκες και τους στόχους μας. Πέραν όμως των μέτρων αυτών, φάνηκε ότι είναι και ισχυρό μέτρο που μπορεί να αντιμετωπίσει συγκεκριμένα οικονομικά προβλήματα και είχε και ένα άλλο πολύ σημαντικό επίτευγμα, το ότι έδειξε πόσο αποτελεσματικά είναι τα κοινοτικά θεσμικά όργανα στην αντιμετώπιση των προκλήσεων της οικονομικής κρίσης. Και μάλιστα μια στιγμή που αυτή η αντίδραση ήταν πολύ σημαντική. Κατάφεραν λοιπόν τα διαρθρωτικά ταμεία να βοηθήσουν στην αποκατάσταση της εμπιστοσύνης ε, ως προς τη δυνατότητα αντίδρασης της Ένωσης στην κρίση. Οπότε, κατά τη γνώμη μου, αυτή ήταν πολύ σημαντική η εμπειρία που αποκομίσαμε από την μετατροπή και την ελαστικότητα των διαρθρωτικών ταμείων. Τροποποιήθηκαν λοιπόν τα μέσα συνοχή για να αντιμετωπιστεί καλύτερα η κρίση και επίση ανταποκρίθηκαν σε μια γενικευμένη απέτηση την ανάγκη απλούστευσης ε, της ε, διαχείρισής του σε όλες τις φάσεις και στη φάση της προετοιμασίας των προγραμμάτων αλλά και στη φάση επαναπροσανατολισμού των προτεραιοτήτων και αντιμετώπισης βραχυπρόθεσμων προβλημάτων. Έτσι, αξιοποιήθηκαν πολύ καλύτερα τα διαρθρωτικά ταμεία, χάρη σε αυτή την ευελιξία. Και ελπίζω πολλές από τις μεταρρυθμίσεις που έγιναν και από τις αλλαγές να διατηρηθούν και στο μέλλον. Αγαπητοί συνάδελφοι, νομίζω ότι όλοι έχουμε επίγνωση της κρισιμότητας της στιγμής. Και οι προτεραιότητες μας αυτή την κρίσιμη στιγμή είναι η ανάκαμψη και η δημιουργία νέων ευκαιριών, διαφυλάσσοντας το κοινωνικό μας μοντέλο. Έχουμε ένα ανεκτήμητο εργαλείο, την πολιτική συνοχή στον αγώνα αυτό. Η πολιτική συνοχή έχει αποδείξει ακόμη, ότι ακόμη και στι δυσκολότερε στιγμέ τη κρίση, με αλλαγέ, με ευελιξία και με προσαρμοστικότητα, με σωστό προσανατολισμό, σωστό συντονισμό και με την απαραίτητη διαφάνεια, έχουν μια τεράστια αξία. Αλλά και τεράστιο δυναμικό και ικανότητα να ανταποκριθούν στις προκλήσεις. Και αυτό ήταν ένα πολύ σημαντικό δίδαγμα που αντλήσαμε από την κρίση. Ο προσανατολισμός λοιπόν της πολιτικής συνοχής στις πραγματικές ανάγκες των Ευρωπαίων πολιτών αποτελεί ευθύνη και καθήκον μας και αυτό θα είναι και η σημαντικότερη συμβολή μας στη διακυβέρνηση. Ευχαριστώ. Euh, Ευχαριστώ αγαπητοί συνάδελφοι, κύριε Γερουσιαστή. Βλέπουμε λοιπόν καλύτερα πώς χρησιμοποίησε η Ισπανία τα διαθέσιμα κονδύλια για να ασκήσει μια πολιτική εξαιρετικά θαραλέα που αρχίζει να αποφέρει καρπούς, ιδιαίτερα στο εξωτερικό εμπόριο που τα αποτελέσματα είναι εντυπωσιακά. Κάποιος καρπούς επίσης ε, αποφέρει την ανεργία που παραμένει το πρόβλημα υπαριθμών ένα στη χώρα σας. Αλλά είναι σαφές πως οι προσπάθειες που έχουν καταβληθεί στη χώρα τις οποίες οι γερουσιαστές ε, εκφράστηκαν θα πρέπει να χρησιμεύσουν ως παράδειγμα για τις υπόλοιπες χώρες συμπεριλαμβανομένες και της δικής μου. Να δώσω τώρα το λόγο στην τελευταία ομιλητρία του πάνελ, την κυρία Μπερούτε Τεβεσάιτ, που αντιπροσωπεύει το Κοινοβούλιο της Λιθουανίας που μάλιστα είχε την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη διάρκεια του δεύτερου εξαμήνου του 2013 και με την οποία κλείσαμε τις διαπραγματεύσεις μετά από την Ιρλανδία και με τη Λιθουανία τη διαπραγματεύσει όχι μόνο για τον Ευρωπαϊκό Προπολογισμό του 2014 αλλά και για το σύνολο του Δημοσιονομικού Πλαισίου 2014-2020. Έχετε το λόγο κυρία μου. Ε, σας ευχαριστώ, εκπρόσωποι των Εθνικών Κοινοβουλίων ε, και ε, ε, κυρίες και κύριοι. Είμαστε ευτυχείς με την έκβαση της Λιθανικής Προεδρίας στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Έχουμε κάνει ό,τι είχαμε προγραμματίσει και μάλιστα πολύ περισσότερο. Γι' αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους σας για τη συνεργασία σας και να ευχηθώ κάθε επιτυχία στην Ελλάδα που ανέλαβε τα ενία από εμά. Η σημερινή εβδομάδα στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου είναι μια εξαιρετική ευκαιρία για να μπορέσουμε να αναπτύξουμε τον πολιτικό διάλογο καθώς ε, προσπαθούμε να ε, ε, φτιάξουμε την ευρωπαϊκή οικονομία και την ευρωπαϊκή ανάπτυξη. Είναι απαραίτητο τα εθνικά κοινοβούλια να συμμετέχουν ενεργά στις διαδικασίες ε, και του ευρωπαϊκού εξαμήνου, γιατί με αυτόν τον τρόπο συμβάλλουν στον δημοκρατική νομιμότητα. Ε, με τα χαρά θα μοιραστώ μαζί σας τις καλές πρακτικές της Λιθουανίας. Σήμερα θα μιλήσω για τον αντίκτυπο της ευρωπαϊκής διευθυντικής βοήθειας για την ανάκαμψη της οικονομίας μας και το χειρισμό των συνεπειών της κρίσης. Όσον αφορά την απορρόφηση της ε, ευρωπαϊκής βοήθειας σε ολόκληρη την Ένωση, την τελευταία χρηματοδοτική περίοδο βλέπετε ότι η Λιθουανία βρίσκεται στο πάνω κομμάτι της κλίμακας και ε, ανάμεσα στους πρωτοπόρους. Όσον αφορά την Ευρωπαϊκή διεθνική Βοήθεια για τη Λιθουανία, αυτή ανήλθε στο, στα 6,7 δις ευρώ. Πάνω από το 14% επενδύθηκε στην ανάπτυξη των ανθρωπίνων πόρων. Το μεγαλύτερο κομμάτι ε, της, του συνόλου της ευρωπαϊκής χρηματοδότησης επενδύθηκε στην οικονομική ανάπτυξη και πάνω από το 39% στην πρόθεση της συνοχής, δηλαδή περιβάλλον, τοπική ε, χορταξική υποδομή και το ε, πρόθεση του τουρισμού, η βελτίωση των δημοσίων υπηρεσιών, ε, παιδεία, υγεία. Ποια είναι τώρα η κατάσταση της εφαρμογής όσον αφορά τα επιχειρησιακά προγράμματα. Στις περισσότερες περιπτώσεις, σχεδόν όλα τα κονδύλια της Ευρωπαϊκής Διαθετικής Στήριξης ε, διανεμήθηκαν για τα προγράμματα. Αυτό σημαίνει πως δεν έχει υπάρξει καθυστέρηση. Η Ευρωπαϊκή Διευθυντική Βοήθεια χρησιμοποιήθηκε για την αναζωογόνηση της οικονομίας της Λιθουανίας και της Ένωσης βεβαίως. Ε, η κατάσταση και οι διαδικασίες αναθεωρήθηκαν ούτως ώστε να μειωθεί το αίτημα για, τρέχους, για ρευστότητα μέσα στο πρόγραμμα της ε, εφαρμογής. Αυξήθηκε η χρηματοδότηση για τα δημοσιονομικά μέσα, αλλά αυξήθηκε και η χρηματοδότηση για τις, ε, τους τομείς προτεραιότητας. Φυσικά, η εξοικονόμηση ενέργειας στα ιδιωτικά αλλά και στα δημόσια κτίρια, η μόνωση αυτών ε, ήταν πολύ σημαντική προτεραιότητα. Η μετάβαση από τα παραδοσιακά καύσιμα στα ανανεώσιμα πολύ σημαντική επίσης, ιδιαίτερα όσον αφορά τη βιομάζα, η πρόθεση των τεχνολογιών που βασίζονται στην ε, καινοτομία και στην έρευνα και στην ανάπτυξη, αλλά και η περιφερειακή ανάπτυξη ήταν ανάμεσα στους στόχους μας, διότι συμφωνώ απολύτως με τον Γενικό Διευθυντή ότι Υπάρχει αυξανόμενη διαφορά, ανισότητα ανάμεσα στις μεγάλες πόλεις και τις περιφέρειες εντός των κρατών αλλά και στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης, επιπλέον μέτρα ελήφθησαν για να αυξηθεί η απασχόληση χρησιμοποιήσαμε προνομιακά δάνεια, συνδυασμό μέτρων ε, δημοσιονομικών με ε, ε, επιδοτήσεις, χρηματοδοτήσαμε μέτρα δραστήρια για την αγορά εργασίας, αν και έχουμε μεγάλη ανεργία που έχει ξεπεράσει το 10%. Έχουμε, εξακολουθούμε να έχουμε διαρθρωτική ανεργία, διότι οι ανάγκες της αγοράς εργασίας δεν καλύπτονται από ειδικευμένους εργαζόμενους. Οπότε τώρα, αντίκτυπος στην οικονομία της Λιθουανίας. Η το ετήσιο ποσοστό αύξησης του ΑΕΠ μας είναι 1,57 ψηλότερο για την περίοδο 2004 με 2013. Αυτό σημαίνει δηλαδή λίγο ψηλότερο από το μέσο όρο της Ένωσης. Κάθε λίτας που επενδύεται αποδίδει δύο σχεδόν λίτας όσον αφορά την αύξηση του ονομαστικού ΑΕΠ. Και η, το ποσοστό ανεργίας προβλέπεται να είναι 4,6% χαμηλότερο. Επιπλέον όθηση δίνεται από τα δημοσιονομικά μέσα που διευκολύνουν τη μείωση του κόστους των επενδύσεων και έμεσα πολλαπλασιάζουν την αξία των ιδιωτικών επενδύσεων. Λόγω της ε, δημοσιονομικής, ε, μάλλον της χρηματοπιστωτικής κρίσης, τα κονδύλια του Κοινωνικού Ταμείου χρησιμοποιήθηκαν ώστε να βλύνουν τα αποτελέσματα, τις επιπτώσει μάλλον της κρίσης, γιατί προορίστηκαν στα θέματα της ανεργίας. Τομίζω που οι πολίτες μας ε, βλέπουν περισσότερο τα ωφέλη της χρηματοδότησης από την Ένωση. η μελέτη που έγινε το 2013 για το πώς αντιλαμβάνεται ο κόσμος τον αντίκτυπο των ευρωπαϊκών κονδυλίων έδειξε ότι το 58% των συμμετεχόντων νιώθουν τη βελτίωση στον τομέα των μεταφορών και στις υποδομές. Το 33% είδε τα ωφέλη των ευρωπαϊκών κονδυλίων στον τομέα της παιδείας και 17% πιστεύει ότι ο τομέας του περιβάλλοντος ωφελήθηκε περισσότερο. Μόνο 2% από τους ερωτώμενους αισθάνθηκαν τα ωφέλη των ευρωπαϊκών κονδυλίων στον τομέα της δημόσιας διοίκησης. What main factors Ποιοι είναι οι βασικοί παράγοντες της αποτελεσματικής χρήσης των ευρωπαϊκών κονδυλίων. Καταρχήν, κεντρικό και διαχείριση και σύστημα ελέγχου για όλα τα επιχειρησιακά προγράμματα μία και μόνη αρχή διαχείρισης. Σαφής χωρισμός ε, κατανομή μάλλον ευθυνών. Μικρές αλλαγές στις ε, θεσμικές ρυθμίσεις σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο, διατηρώντας όμως ε, τους έμπειρους συνεργάτες και τυποποιημένοι κοινοί κανόνες και διαδικασίες. Επίσης, η προετοιμασία των ε, προγραμμάτων, δηλαδή έγκαιρη προετοιμασία των εθνικών στατηγικών εγγράφων για την ε, στρατηγικό σχεδιασμό των επενδύσεων, αλλά και έγκαιρη προετοιμασία προγραμμάτων από τους ίδιους τους δικαιούχους. Όλα αυτά είναι τεράστια σημασία. Of administrative procedures η απλοποίηση των διοικητικών διαδικασιών. Πιο ευέλικτε μέθοδοι ε, πληρωμών, αξιολόγηση των προγραμμάτων και επιλογής αυτών, η σμίκρινση των, της διαδικασίας επαλήθευσης ε, και ελέγχου των αιτήσεων για τα προγράμματα, επίσης ε, η χρήση των πληρωμών με ένα απλοποιημένη, με απλοποιημένη βάση κόστου, δηλαδή κατά ποσέ και συγκεκριμένα κόστη ε, μοναδιαία. Η χρήση ε, δημοσιονομικών μέσων επίσης, ε, δηλαδή η δυνατότητα ε, αποπληρωμής μεγάλης μόχλευσης με βάση αυτών, ε, αυτά τα κονδύλια, καθώς και η χρήση των συστημάτων πληροφορικής που χρησιμοποιούνται σε όλες τις τυποποιημένες καθημερινές διαδικασίες και είναι ένα καθημερινό εργαλείο για τη διαχείριση των ευρωπαϊκών κονδυλίων. Ποια είναι τα διδάγματα που αποκομίσαμε τώρα, οι κίνδυνοι ποιοι είναι. Η καθυστερημένη ε, εφαρμογή σημαίνει αυξημένους κινδύνους στο τέλος της ε, προγραμματικής περίοδου και επίσης άλλος κίνδυνος είναι το να, μην, το να μην υπάρχει μια ολοκληρωμένη εθνική τομεακή στρατηγική. Αυτό σημαίνει καθυστέρηση στην έναρξη των προγραμμάτων. Ποιες είναι οι πιθανέ λύσεις. Καταρχήν μεταβατικές διαδικασίες οι οποίες θα έχουν εγκριθεί. Οι, προηγούμε, προϋποθέσεις για την έγκριση των στρατηγικών προγραμμάτων δράσης και η βελτίωση των διαδικασιών για τις κρατικές προμήθειες που κάποιες φορές είναι ο βασικός λόγος καθυστέρησης των προγραμμάτων. Κύριες αρχές για τη διαχείριση και το σύστημα ελέγχου. Η ε, διαδοχή, η οτυποποίηση των διαδικασιών, η απλοποίηση των, της διαδικασίας ή των απαιτήσεων. Αυτό είναι ένα θέμα για την, ε, ε, για την Επιτροπή και η χρησιμοποίηση των εργαλείων ε, της πληροφορικής. Ποια είναι τώρα τα επιτεύγματα. Η Τα ευρωπαϊκά διευθυντικά ταμεία συνέβαλαν σημαντικά στην οικονομική και κοινωνική πρόοδο στη Λιθουανία σε πολλούς τομείς. Αυτή τη στιγμή πολλά σημαντικά αποτελέσματα έχουν ήδη επιτευχθεί χάρη στα ευρωπαϊκά κονδύλια. Πάνω από 170.000 άνεργοι οι ε, άνθρωποι που ήταν υπό την απειλή της ανεργίας συμμετείχαν σε προγράμματα ε, ε, κατάρτισης, σχεδόν 40.000 άνεργοι καταρτίστηκαν επαγγελματικά. 2.500 επιδοτήσεις για ερευνητικές επιστημονικές δραστηριότητες δόθηκαν, χορηγήθηκαν σε φοιτητές, επιστήμονες και ερευνητές. Πάνω από 2.500 επιχειρήσεις ωφελήθηκαν από επενδύσεις για καινοτομία, από χρηματοπιστωτική βοήθεια που δόθηκε για 5,8 χιλιάδες μικρομεσαίες επιχειρήσεις. 1,5, μάλλον 1.500 χιλιόμετρα ε, οδών αποκαταστάθηκαν ή κατασκευάστηκαν. 775 πόλεις και χωριά συνδέθηκαν ε, με βριζονικό ίντερνετ. Ανακαινίστηκαν 769 κτίρια του δημόσιου τομέα, όπως σχολεία, νηπιακή σταθμή, νοσοκομεία και ούτω καθεξής. και πάνω από 700.000 καταναλωτές ωφελήθηκαν από την αυξημένη ποιότητα και την αξιοπιστία της παροχής ενέργειας και βέβαια χαμηλότερους λογαριασμούς θέρμανσης. Πολύ σημαντικό αυτό το στοιχείο. Τα δίκτυα ίδρευσης και αποχέτευσης επίσης ανακαινίστηκαν ενώ κατασκευάστηκαν νέα σε 237 περιοχές. Έκλεισαν 242 χωματερές ή ε, καθαρίστηκαν, εξηγιάνθηκαν. Ε, επίσης, ε, η οικονομία χαμηλής ε, προστιθέμενης αξίας μετατράπει σε οικονομία υψηλής προστιθέμενης αξίας και αυτό ήταν πολύ σημαντικό. Άρα λοιπόν να σας πω τώρα ποιοι είναι οι βασικοί μας στόχοι για το μέλλον. Η ευφυής και καθολική ανάπτυξη, περαιτέρω προώθηση της έρευνας και της καινοτομίας, βελτίωση της ποιότητας της παιδείας, αποδοτικότητα της δημόσιας διοίκησης και ανάπτυξη της ψηφιακής κοινωνίας. Δεύτερον, η βιώσιμη ανάπτυξη Δηλαδή, η ανάπτυξη σύγχρονων βασικών υποδομών, καλύτερο περιβάλλον για τις επιχειρήσεις, καθώς και βιώσιμη και αποτελεσματική χρήση των φυσικών πόρων και σημείο η ασφάλεια και η, η υπηκότητα, δηλαδή η βελτίωση της απασχόλησης, η μείωση της στόχης, του κοινωνικού αποκλεισμού και συνδυασμός όλων αυτών με κοινωνική και εδαφική συνοχή. Συμφωνώ με την Κομισιόν ότι η επένδυση των ευρωπαϊκών ε, τα κονδυλίων θα πρέπει να προσανατολίζεται στα αποτελέσματα που θα πρέπει να είναι περισσότερες και καλύτερες θέσεις απασχόλησης για τους πολίτες μας. Σας ευχαριστώ. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ, ε, κυρία Γερουσιαστά. Συγχαρητήρια για τις προσπάθειες της Λιθουανίας που ε, προσεχώς ε, πρόκειται να γίνει μέλος ε, από ό,τι φαίνεται της ζώνης του ευρώ. Λοιπόν, διάφοροι κοινοβουλευτικοί έχουν ζητήσει το λόγο. Θα δώσω πρώτα το λόγο στον κύριο Κρότμανής γιατί πρέπει να πάει και σε μια άλλη συνεδρίαση. Ναι, ναι, πρέπει να πάω στη Ρέγγι. Γι' αυτό κάποιοι δεν είναι παρόντες. Θα ήθελα ε, να προσέξετε κάπως αυτά που θα πω και κυρίως ε, προς τη Γενική Διεύθυνση. Πρέπει αυτή η συνάντηση να αντιμετωπίσει τα πραγματικά προβλήματα. Μέχρι στιγμής έχουμε ακούσει καθόλου προβλήματα. Πολύ ωραία προοπτική για το μέλλον, πολύ καλές ε, παρουσιάσεις από την Ελλάδα και την Λιθουανία. Αλλά υπάρχουν πολλά προβλήματα και θα προσπαθήσω να τα αναφέρω τι σχέση έχει η Επιτροπή Προϋπολογισμών και τα Ταμεία Συνοχής. Αυτό το πρόβλημα, ο ρόλος. Θέλουμε να αυξηθούν οι πληρωμές. Α, αυτό που μας ενδιαφέρει περισσότερο είναι το resta liquide, αυτό που ακόμη δεν έχουν εκταμιευθεί. Αλλά οι αντίπαλοι μας, που μας έδωσαν μόνο 906 εκατομμύρια. Χρησιμοποιούν αυτό το όργανο, το Uresta Liquide, που είναι πάνω από 200 δισεκατομμύρια, που δεν έχουν εκταμιευθεί. Και 70% από αυτά είναι πόροι συνοχής. Και το ερώτημα λοιπόν είναι, μπορούμε να το υπερβούμε αυτό. Είναι μεγάλο πρόβλημα. Τελευταία φορά στο Στρασβούργο, όταν ε, ε, ψηφίσαμε για τα διάφορα ταμεία είπα να βάλουμε η Ρέγκη να είναι υπεύθυνη για την ε, εκτέλεση των ταμείων. Ε, πρέπει να την ε, αποσύρω γιατί εξεφράστη ζήλια από την Επιτροπή Απασχόλησης και άλλες, οπότε τα επόμενα 7 χρόνια τι θα προκύψει. Κανείς δεν θα είναι υπεύθυνο για την επίβλεψη της εκτέλεσης. Ούτε ακόμη και λογιστικά γιατί είναι τόσο σημαντικό αυτό. Θα σας δώσω στοιχεία που ίσως να μην ξέρετε. Τα τελευταία στοιχεία, επίσημα, 1η Δεκεμβρίου 13 για την 1η Ιανουαρίου δεν έχουμε. Να δούμε τι είναι αυτά τα ραλ, τα υπόλοιπα προς ακαθάριση δηλαδή, και γιατί δεν μειώνονται. Και τώρα δεν θα ε, εφαρμόσω την πολιτική της Κομισιόν που δεν θέλει να δείξει με το δάχτυλο κανένα γιατί εδώ ε, έχουμε προσώπους από διάφορες χώρες που θέλουν να ξέρουν τα πάω καλά από πλευράς απορρόφησης, τα πάω καλά από πλευράς απορρόφησης του Κοινωνικού Ταμείου, του Περιφερειακού Ταμείου, ποια είναι τα αποτελέσματα. Το κύριο πρόβλημα του υπόλοιπου προς ε, καθάριση είναι ότι αν πάρουμε μαζί το κοινωνικό και το περιφερειακό 16% ε, είναι 60% μόνο η απορρόφηση. Το 40% λοιπόν της προηγούμενης προγραμματικής περίοδου ε, δεν έχουν εκταμιευθεί και 16 χώρες είναι κάτω από το μέσο όρο και η διαφορά ανάμεσα στην καλύτερη χώρα που είναι η Λιθουανία και τη χειρότερη που είναι η Ρουμανία είναι 216%. Και πρέπει να πω ότι αν εξετάσουμε τις χώρες που αντιμετωπίζουν πραγματική κρίση, πρέπει να πούμε ότι η Ελλάδα τα πάει καλά. Με 71%. Πολύ καλά. Πολύ καλά. Είναι μέσα στους πρώτους πέντε. Το ίδιο ισχύει για την Ισπανία. Είναι στην ενδέκατη η θέση. 62%. Λίγο πάνω από το μέσο όρο. Αλλά αν εξετάσετε τη χειρότερη κατάσταση, θα διαπιστώσετε ότι η Ρουμανία και η Βουλγαρία που εντάχθηκαν το 2007 δεν επέτυχαν μέσα σε 7 χρόνια να εφαρμόσουν, ε, να απορροφήσουν αρκετά. Η Ρουμανία είναι πολύ πίσω. Είπαμε 2,5% δηλαδή 2,5 φορές κάτω από τον καλύτερο. Κανείς δεν έχει κάνει ανάλυση ούτε στην Επιτροπή Περιφερειακών Υποθέσεων γιατί είναι έτσι τα πράγματα, γιατί έχουν προβλήματα αυτές οι χώρες. Και δεν αφορά μόνο αυτές τις δύο τελευταίες χώρες που δεν είναι πια και τόσο πρόσφατες. Ε, θα δείτε και ότι η Ιταλία για παράδειγμα είναι στην 26η θέση. 45% απορρόφηση των πόρων συνοχής και του Περιφερειακού Ταμείου. Και η Κροατία 24η θέση, 48%. Και η Αυστρία που δεν παίρνει πολλές χρηματοδοτήσεις, αλλά είναι μόνο στην 23η θέση. Κανείς λοιπόν, επειδή καμία επιτροπή δεν είναι αρμόδια, κανείς δεν έχει αναλύσει. Θα ζητούσα λοιπόν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, παρακαλώ αλλάξτε πολιτική, ελάτε στην Περιφερειακή Επιτροπή, στην Επιτροπή Προπολογισμών, εξηγήστε γιατί υπάρχουν αυτά τα προβλήματα και να δείξετε με το δάχτυλο ποιοι φταίνε γιατί αν δεν ε, βελτιωθεί η κατάσταση θα ε, οξυνθεί το πρόβλημα. Και για το κοινωνικό ταμείο είναι ακόμη χειρότερη η κατάσταση. Και δεν τα πάνε τόσο καλά η Ισπανία και η Ελλάδα. Όταν είναι τόσο ψηλή η ανεργία, άμα δείτε πώς έχουν απορροφήσει ε, κοινωνικούς πόρους, η Ισπανία είναι λίγο κάτω από το μέσο όρο και η Ελλάδα το ίδιο. και επίσης η Σλοβακία, η Κύπρος, η Ουγγαρία, ακόμη και η Γαλλία. Είναι στην 20η θέση η Γαλλία, όχι τόσο καλά. Και είναι θέματα καταπολέμησης της ανεργίας. Και πάλι η καλύτερη από τη χειρότερη είναι 2,5 φορές η διαφορά. Και 6% είναι κάτω από τον μέσο όρο απορρόφησης που είναι 64%. Και αυτά είναι εύκολοι πόροι. Είναι εύκολα προγράμματα. Δεν χρειάζονται υποδομές κτλ. Και κάτι τώρα για τη Γενική Διεύθυνση της Κομισιόν. Αν δεν υπάρχουν ε, επισήμως ε, επιτροπές ε, επιτήρησης, δεν είναι δυνατόν όλοι να είναι υπεύθυνοι. Σας παρακαλώ, ε, ανασκουμποθείτε, δώστε γνώμη. Δεν το έχετε κάνει μέχρι στιγμής. Με συγχωρείτε. Πολύ γενικόλογα. Θέλουμε συγκεκριμένα αναπρόβλημα. Γιατί συμβαίνει αυτό. Δεύτερον, νέες δραστηριότητες. Τελειώνω, τελειώνω. Ναι, υπάρχουν πάρα πολλοί ομιλητέ που έχουν το λόγο. Παρακαλώ, τελειώνετε. Εντάξει, θα τελειώσω. Ευχαριστώ πολύ και με συγχωρείτε, λέει ο πρόεδρο. Αντριέλ Γκαλαζεύσκη, του Πολωνικού Κοινοβουλίου. Παρακαλώ. Αγαπητέ συνάδελφοι, παρακαλώ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πολωνία αξιοποιεί τα ευρωπαϊκά κονδύλια. Και μάλιστα έχουμε, θα έπρεπε να έχουμε καλύτερη ε, σύνδεση του Υπουργείου Υποδομών ε, ε, έχουμε καλύτερη σύνδεση μεταξύ των δύο Υπουργών Υποδομών και ε, ανάπτυξης και μάλιστα είναι και αντιπρόεδρος της κυβέρνησης ο αρμόδιος υπουργός. Κάτι που δείχνει πόση μεγάλη σημασία αποδίδουμε και πόσο θα αξιοποιούμε τα ευρωπαϊκά κονδύλια. Επίσης η εκταμείευση των κονδυλίων και η σωστή αξιοποίησή τους είναι πολύ σημαντική. Ακόμη πιο σημαντική όμως είναι η ορθή, ο ορθός προσδιορισμός των στόχων που θα πρέπει να εξυπηρετούν αυτά τα κονδύλια. Ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είπε ότι θέλουμε ένα προσανατολισμό προς τα αποτελέσματα. Αυτό κανονικά πρέπει να είναι αυτονόητο. Εγώ είμαι πολλά χρόνια στη δημόσια διοίκηση και ανέκαθεν όταν αξιοποιήσαμε κονδύλια στη δημόσια διοίκηση ήμασταν προσανατολισμένοι προς τους στόχους. Εννοείται προς τα αποτελέσματα. Και είναι περίεργο που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τώρα το αντιλήφθηκε ότι θα πρέπει να είναι προσανατολισμένη προς τα αποτελέσματα και τους στόχους. Είναι πολύ σημαντική λοιπόν η στόχη, γιατί μερικές φορές τελείως ασυλλόγιστα δαπανούμε υψηλά κονδύλια και δημιουργείται μια παθολογική κατάσταση. Για παράδειγμα, είχαμε ανελαστική δαπάνη πολλών κονδυλίων σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αυτό δημιουργεί ε, παθολογικές καταστάσεις και διαφθορά σε μια χώρα μέλος. Επίσης υπήρχαν διαταραχές ε, στο, στην λειτουργία του ενεργειακού συστήματος και μειώθηκε η ενεργειακή απόδοση σημαντικών πηγών ενέργειας που αποτελούν τη βάση της ενεργειακής ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα ήθελα λοιπόν να παροτρύνω και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη-μέλη να μην εμένουν δογματικά σε συγκεκριμένε ε, λύσεις. θα έλεγα περισσότερο να προσανατολίζονται και να κατευθύνονται από την κοινή λογική ε, όταν ε, αξιοποιούν τα κονδύλια. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κύριε συνάδελφε. Θα ήθελα τώρα να δώσω το λόγο στον κύριο Καριέλο από την ε, Ιταλική Βουλή. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είναι πολύ σημαντικό να μιλήσουμε σήμερα για την αιρεσιμότητα στη χρήση των επενδύσεων. Με τη δημιουργία του ενιαίου νομίσματος, όλα τα κράτη-μέλη εκχωρήσαμε την αυτονομία και το τη δυνατότητα νομισματικών ελιγμών και μάλιστα πέραν της εκχώρησης αυτής αναλάβαμε μια σειρά δημοσιονομικών υποχρεώσεων που ανάγκασαν τα κράτη-μέλη να αυξήσουν τα έσοδα και να μειώσουν τις δαπάνες τους. Τώρα, εξαρτούμε τις επενδύσεις από τη λήψη συγκεκριμένων μέτρων οικονομικής πολιτικής που λαμβάνει το Συμβούλιο. Αυτή η μακροοικονομική αιρεσιμότητα δημιουργεί πολλά προβλήματα γιατί περιορίζει τις δυνατότητες ενός κράτους μέλους να προβεί σε επενδύσεις. Και μάλιστα πλήγει περισσότερο τις χώρες που έχουν τα μεγαλύτερα προβλήματα για να τηρήσουν το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Η πρόταση μας λοιπόν θα ήταν μια αναθεώρηση των ε, τριών κορυφών και πλευρών του τριγώνου που μας παρουσίασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και θα πρότεινα να αντικαταστήσουμε την εξηγία στη δημοσιονομική, τη δημοσιονομική πολιτική από την επενδυτική πολιτική. Θα πρέπει οι επενδύσεις να, στη, να προωθούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και να χρηματοδοτούνται άνεφόρων. Γιατί πάνω απ' όλα είμαστε μία κοινότητα, μία ένωση. Θα πρέπει λοιπόν να έχουμε εμπιστοσύνη σε όλα τα μέλη αυτής της ένωσης. Επίσης, το Συμβούλιο θα πρέπει να θεσπίσει μία πολιτική που θα ενισχύει τις επενδύσεις, θα τις προωθεί και θα επαναφέρει στα κράτη-μέλη χάρη σε επενδύσεις τη δυνατότητα να τονώσει την οικονομία. Μια δυνατότητα που την έχασαν με την υπογραφή του Συμφώνου σταθερότητα και Ανάπτυξης. Επίσης, τα χρησιμοποίητα ε, διαφθορτικά κονδύλια δημιουργούν πρόβλημα εξαιτία τη αδυναμίας των ε, κρατών μελών να συγχρηματοδοτήσουν. Γιατί έχουν μία επιπλέον υποχρέωση εκεί με τη συγχρηματοδότηση. Πώς πιστεύετε ή πώς απαιτείται από μία χώρα να δώσει κίνητρα για τις επενδύσεις αν ε, δεν έχει πια τη δυνατότητα να αποφασίζει για την οικονομική της πολιτική. Στερηθήκαμε το δικαίωμα χάραξης οικονομικής πολιτικής. Θα πρέπει ως αντιστάθμισμα να λάβουμε αν μη τι άλλο την ε, προώθηση των επενδύσεων ανεφόρων και χωρίς αυτή την αιρεσιμότητα που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Επίσης ήθελα να πω ότι η Ιταλία κατάφερε να εκταμιεύσει πολλά κονδύλια και να εθετήσει το 53% των στόχων. 48% ήταν το αρχικό ποσοστό, η πρόβλεψη για το ποσοστό εκταμίευσης και εμείς ξεπεράσαμε αυτό το στόχο. Φτάσαμε στο 53%. Στο μέλλον όμως περιμένουμε και από το Συμβούλιο μία χειρονομία προκειμένου να, γίνονται επενδύσει χωρίς υπερβολική αρεσιμότητα. Η κυρία Χέλγα Τρίπελ έχει το λόγο από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Να επανέλθω σε αυτά που είπε ο Γενικό Διευθυντή. Είπε σήμερα το πρωί ότι τα προγράμματα πρέπει να είναι στρατηγικά. Νομίζω ότι χρειάζεται μια πολύ στρατηγική προσέγγιση. Ε, θα οδηγούσε στο να αποσυνδέσουμε την ανάπτυξη από τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα. Αλλά αναφέρθηκαν προγράμματα εξοικονομήσεων ενέργειας και το πέρασμα από τα ορυκτά στα ανανεώσιμα κάψιμα. Αλλά θα έπρεπε στο κέντρο της προσέγγισης μας ε, να υπάρχει προσπάθεια να λαμβάνουμε υπόψη την ανάγκη μείωσης ε, των ε, εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα και προώθηση των ανανεωσίμων. Όταν συζητάμε για αυτοκινητοδρόμους, για παράδειγμα, συζητήθηκε αν αυτή θα είναι η στρατηγική μας προσέγγιση. Ο καλύτερος τρόπος να αναπτύξουμε ε, την οικονομία μας είναι να συνδυάσουμε την ανάπτυξη με τη μείωση των εκπομπών. Ευχαριστώ πολύ, Χέλγα, λέει ο πρόεδρος, ο Ιβάιλο Κάλφιν, μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ευχαριστώ, πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, ευχαριστώ πολύ όλους τους ε, συναδέλφους από τα Εθνικά Κοινοβούλια για την παρουσία τους γιατί πρέπει να συζητήσουμε και να συντονίσουμε τις προσπάθειες μας στο μέλλον. Θα εστιάσω σε λίγα θέματα που θα συζητηθούν τους προσεχείς μήνες και όπου η συνεργασία μεταξύ Εθνικών και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και η ε, συμφωνία είναι ε, αναγκαία. Σχετίζονται γενικότερα με τον προπολογισμό της Ένωσης. Το πρώτο θέμα αφορά την ευελιξία του προϋπολογισμού. Ξέρετε ότι για πρώτη φορά εγκρίναμε μειωμένο, μειωμένους καλύτερα προϋπολογισμούς για την περίοδο μέχρι το 2020 και συμφώνησε το Κοινοβούλιο, το Ευρωπαϊκό γι' αυτό, γιατί εισήχθησαν στοιχεία περισσότερης ε, ευελιξίας. Μία θα είναι η ενδιάμεση αναθεώρηση. Ελπίζουμε η οικονομική συγκυρία να βελτιωθεί και γι' αυτό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επιμένει και είναι στην Διοργανική Συμφωνία να υπάρχει μία πλήρης ενδιάμεση αναθεώρηση του ενωσιακού προϋπολογισμού το 2016. Δηλαδή, η διαδικασία αυτή θα πρέπει να γίνει αυτή η αναθεώρηση. Και εδώ θα πρέπει να παίξουν το ρόλο τους και τα εθνικά κοινοβούλια. Θα έχουμε καλύτερη ιδέα για το τι θα γίνει μέχρι το 2020, το 2016. Το 2016 θα καταλαβαίνουμε καλύτερα, θα έχουμε μια καλύτερη ιδέα για το τι θα γίνει μέχρι το 2020 στις εθνικές οικονομίες και θα έχουμε ένα νέο κοινοβούλιο και μια νέα επιτροπή. οι εθνικές κυβερνήσεις ε, μπορεί βέβαια να είναι κάπως απρόθυμες όπως και στο παρελθόν να γίνει αυτή η μεσοπρόθεσμη ή ενδιάμεση αναθεώρηση. Οπότε θα ήθελα ε, να μας στηρίξουν τα Εθνικά Κοινοβούλια για να υπάρξει αυτή η διαδικασία. Δεύτερο θέμα. Μια ιδιαιτερότητα του ενωσιακού προπολογισμού που δεν έχουμε ποτέ συζητήσει. Οι ίδιοι πόροι. Ο ενωσιακός προπολογισμό ε, χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους και από ίδιους πόρους. Κατά 80% ωστόσο χρηματοδοτείται από εθνικές συνεισφορές και μόνο κατά 20% από γνήσιους ίδιους πόρους. Αυτή δεν ήταν η αντίληψη των συνθήκων. Οι συνθήκες ε, είχαν τη γενικότερη προσέγγιση ότι ο ενωσιακός προπολογισμό θα πρέπει να είναι πολύ πιο ανεξάρτητος και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θέτει το θέμα των ίδιων πόρων αλλά δεν το θέτει για να αυξηθεί ο ενωσιακός προπολογισμό, αλλά για να γίνει πιο ανεξάρτητος και για να βελτιωθεί και η κατάσταση των εθνικών προϋπολογισμών, διότι φυσικά οι εθνικές συνεισφορές αυξάνουν ε, τα ελλείμματα των εθνικών προϋπολογισμών και όλες τις άλλες επιπτώσεις που συζητάμε εδώ στο Ευρωπαϊκό Εξάμεινο. Αν συμφωνήσουμε λοιπόν αυτό το ποσοστό των εθνικών συνεισφορών 80% και μόνο 20% να αλλάξει ας πούμε και να γίνει 60% ήδη υπόρρη και 40% εθνικές συνεισφορές, αυτό θα ελαφρύνει κατά πολύ τους εθνικούς προϋπολογισμούς χωρίς να αυξάνει το σύνολο των ε, δημοσίων δαπανών χωρίς να προστίθενται νέοι φόροι κτλ. Έτσι όμως θα γινόταν πολύ πιο αυτόνομος, πιο προβλέψιμος ο ενωσιακός προπολογισμό και θα απέφευγε ο ευρωπαϊκός προπολογισμό αυτό που κάναμε πέρυσι. Δηλαδή χρειάστηκε να δώσουμε ε, δεκάδες δισεκατομμύρια παραπάνω για να πληρωθούν οι λογαριασμοί της Ευρωπαϊκής Επιτροπής γιατί η δομή και ο τρόπος εκτέλεσης του ευρωπαϊκού προπολογισμού σορεύει αυτό που είπε ο κύριος Γκουτμάνης από τη Λιθουανία, ότι δηλαδή υπάρχουν αυτά τα υπόλοιπα προς εκαθάριση, εναπομένουσες λοιπόν δαπάνες. Πρέπει λοιπόν να πιέσουμε τα κράτη-μέλη και χρειάστηκε να πιέσουμε τα κράτη-μέλη ε, να δώσουν 11 δις για να πληρώσουμε τα ε, απλήρωτα τιμολόγια. Αυτό θα απεφεύγει το αν είχαμε πιο ανεξάρτητο ενωσιακό προπολογισμό. Θα υπάρξει μια υψηλό επίπεδο ομάδα εργασία που θα αρχίσει να εξετάζει τα θέματα αυτά. Το 2016 θα πρέπει να μα έχει υποβάλει διάφορε συναλλακτικέ λύσει. Είναι λεπτό θέμα, αλλά πρέπει να αρχίσουμε να το εξετάζουμε. Και το τελευταίο που θέλω απλώ να αναφέρω. Μια πρόσφατη εξέλιξη που θα χρειαστεί να αντιμετωπιστεί από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο είναι ο προϋπολογισμός ε, για την Ευρωζώνη. Πολύ συχνά οι εθνικές κυβερνήσεις ε, καταλήγουν σε διακυβερνητικές συμφωνίες για το θέμα αυτό. Αλλά αυτό είναι ιδιαίτερα επιζήμιο και για τον προϋπολογισμό της Ένωσης και για το Ευρωπαϊκό Ιδεώδες. Εφόσον από τη μία αποκαλείται ε, ευρωπαϊκός προϋπολογισμός, αλλά από την άλλη αποφασίζεται διακυβερνητικά εκτός των ε, οργάνων της Ένωσης, στην ουσία φύγουμε την ίδια την πορεία της Ευρωπαϊκής ε, Ενοποίησης. Πιστεύω λοιπόν ότι πρέπει και εδώ να μας βοηθήσουν τα Εθνικά Κοινοβούλια ώστε να γίνει τμήμα της κοινοτική μεθόδου και να αποφασίζεται στα πλαίσια της διαδικασίας λήψης αποφάσεων της Ένωσης και όχι μεταξύ κυβερνήσεων. Ευχαριστώ, ευχαριστώ αγαπητέ συνάδελφε, λέει ο Πρόεδρος. Ε, θέλω να επιμείνω σε αυτό το τελευταίο σημείο που ανέφερε ο Ιβάιλο Κάλφιν στις διαπραγματεύσεις μεταξύ Συμβουλίου και Κοινοβουλίου για τις πολιτικές προοπτικές 2014-2020 πολλά κράτη-μέλη επέμειναν ότι ο ευρωπαϊκός προπολογισμός της προσεχούς ε, επταετίας πρέπει να μειωθεί σε σχέση με τον τρέχοντα, δηλαδή του 13 για να ληφθεί υπόψη ότι εφόσον χρηματοδοτείται από τα εθνικά κοινοβούλια, όλοι οι εθνικοί προπολογισμού έχουν υποστεί πολύ σημαντικέ περικοπέ, όπω το εξηγήσω ο Ιβάλλο Κάλφιν. Ω αποτέλεσμα λοιπόν, ο προπολογισμό τη ευρωπαϊκή οικογένεια, ο κοινό μα προπολογισμό, αναγκαστικά έπρεπε και αυτό να περικοπεί. Αλλά ε, είναι πολύ περίεργο να ακούμε τους εκπροσώπους κάποιων κρατών μελών που ήθελαν να μειώσουν τον ευρωπαϊκό προπολογισμό λέγοντας δεν είναι δυνατόν να αυξηθεί η συμβολή μας. Αυτοί οι ίδιοι εκπρόσωποι κρατών μελών θα ήθελαν να δημιουργηθεί ένας νέος κοινό προπολογισμό, αλλά πολύ περιορισμένο, δηλαδή για την Ευρωζώνη. Για ποιο στόχο. Τι διαφορετικό θα εκτελέσει, θα κατορθώσει αυτός ο προπολογισμός και πώς θα χρηματοδοτηθεί. Πώς θα προκύψει. Καμία πολιτική ομάδα, ε, κανείς ε, από τις μεγάλες πολιτικές ε, ομάδες που είναι υπέρ ε, της ευρωπαϊκής ιδέας δεν είναι καταρχήν εχθρικός αυτή την ιδέα, αλλά πρέπει να επιμείνουμε ότι δεν θεωρούμε ότι θα ήταν δυνατόν από τη μία να μην μπορούμε να χρηματοδοτήσουμε τον ευρωπαϊκό προπολογισμό και ω εκ να βρούμε πόρου για τον προπολογισμό αποκλειστικά τη Ευρωζώνη. Αυτό είναι ένα θεμελιώδε πρόβλημα. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο πρέπει να το συζητήσει. Ήδη έγιναν κάποιε τέτοιε συζητήσει ε, στι συναντήσει κορυφή και πιστεύω ότι την κατάλληλη στιγμή, μάλιστα μετά τι ευρωεκλογέ, θα πρέπει να γίνει πολύ πιο συγκεκριμένη συζήτηση γι' αυτό. Και τώρα να δώσω το λόγο στον κύριο Κάζιμιρ Κλέινα από την ε, ε, Πολωνική Γερουσία. Κύριε Γερουσιαστά. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε. Στην Πολωνία θεωρούμε ότι το ευρωπαϊκό εξάμεινο στον επόμενο κύκλο θα αποτελέσει ακόμη πιο αποτελεσματικό όργανο συντονισμού και παρακολούθησης της οικονομικής πολιτικής των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ταυτόχρονα όμως συνειδητοποιούμε ότι οι μεμονωμένες οικονομίες των κρατών μελών ε, είναι πολύ διαφορετικές μεταξύ τους, οπότε αυτός ο συντονισμός θα πρέπει να λάβει υπόψη τις ιδιαιτερότητες των διαφόρων χωρών, ώστε να μην ε, οδηγηθούμε στο αποτέλεσμα η καλή στόχη στόχη όπως είναι η μείωση του διοξιδίου του άνθρακα όπως είπε ο, προ, ο συνάδελφος ε, ε, σε συγκεκριμένες χώρες ε, να έχουν ε, πολλές παρενέργειες και πολύ αρνητικά αποτελέσματα εξαιτίας αυτών των ιδιαιτεροτήτων. Επίσης, τα κράτη-μέλη έχουν και διαφορετικά φορολογικά συστήματα, φορολογικά συστήματα οπότε μια απόπειρα ενοποίησης τους και ομοιογενοποίησης τους ίσω έχει αρνητικά αποτελέσματα σε πολλές χώρες. Η Πολωνία είναι από τους σημαντικότερους αποδέκτες των κοινοτικών κονδύλων και χάρη σε μεγάλο βαθμό και στα κονδύλια αυτά δεν βίωσε τόσο οξία οικονομική κρίση όπως άλλες χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ίσως και γι' αυτό με καλύτερο τρόπο και πολύ πιο καλά αξιοποιήσαμε τα ευρωπαϊκά κονδύλια. Ε, συνειδητοποιούμε όμως ότι και τα κονδύλια αυτά θα έχουν θεμελιώδη σημασία στις επόμενες δημοσιονομικές προπτικές, στην επόμενη δημοσιονομική περίοδο του πολιτού δημοσιονομικού πλαισίου. Ένα σημαντικό πρόβλημα και για την Πολωνία και για άλλε χώρε είναι η ανεργία. Παρόλο που η ανεργία στην Πολωνία δεν είναι τόσο υψηλή όσο στην Ισπανία ή σε άλλε χώρε, παρόλα αυτά είναι οξύτατο πρόβλημα και σε εμά η ανεργία. Ε, αντιμετωπίζουμε και ένα άλλο πρόβλημα που κυρίως ε, ταλανίζει τις νεότερες χώρες μέλη. Στην Πολωνία, για παράδειγμα, έχουμε μαζική έξοδο εργαζομένων προς τις ε, πιο ευημερούσες χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και μάλιστα οι ε, ευημερότερες, ευημερούς αυτές χώρες δεν υποδέχονται ενθουσιοδός τους εργαζόμενους από την Πολωνία από άλλες χώρες, για να το πω κατά θυμισμό. Ε, έτσι έχουμε μία έξοδο εργαζομένων που πολλές φορές είναι πολύ ε, ειδικευμένοι και με πολύ ειδικέ γνώσεις. Αυτή η έξοδος λοιπόν πλήττει και την οικονομία των χωρών προέλευσης. Στην Πολωνία θα επικεντρωθούμε σε σημαντικές επενδύσεις υποδομών. Έχουμε συγκεκριμένη τράπεζα και επίσης επενδυτικούς φορείς που συμβάλλουν στον συντονισμό των πολιτικών για τη χρηματοδότηση σημαντικών έργων υποδομών. Οπότε τα κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα συμβάλλουν και στο μέλλον στην πολύ θετική ανάπτυξη και στη δημιουργία υποδομών στην Πολωνία. Ένα άλλο πολύ σημαντικό στοιχείο είναι η διασυνοριακή συνεργασία. Και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ε, εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης δηλαδή, αλλά και η διασυνοριακή συνεργασία με τις γειτονικές μας χώρες. Στην Πολωνία λαμβάνουμε ιδιαίτερη, ιδιαίτερη υπόψη την κατάσταση στην Ουκρανία, γιατί έχουν πραγματικές τραγωδίες και στο Κίεβο και άλλες, χώρες της, και άλλες πόλεις της Ουκρανίας. Αποδίδουμε ιδιαίτερη προσοχή στη χώρα αυτή. Θα ήθελα να απευθύνω έκκληση προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και στα κρατημέλη να στηρίξουμε την χώρα αυτή, την Ουκρανία, στο δημοκρατικό της δρόμο. Εμεί είμαστε υπέρ τη συνεργασία και κυρίω των επαφών μεταξύ Νέων Πολωνία και Ουκρανία. Είναι δύσκολο βέβαια σε δύο λεπτά να καλύψουμε πολύ περισσότερα θέματα. Σα ευχαριστώ για την προσοχή. Ε, και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Γερουσίστα. Θα δώσω τώρα το λόγο στην κυρία Νόρντεν από το Συνδική Βουλή. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η πολιτική συνοχής είναι ένα πολύ σημαντικό πολιτικό πλαίσιο για την Σουηδία. Και ακόμα και αν οι προοπτικές είναι θετικές, είναι σημαντικό η πολιτική συνοχή να είναι προ όφελο όλων. Εγώ αντιπροσωπεύω μια περιφέρεια στο βόρειο τμήμα τη χώρα μου, όπου η ανεργία των νέων είναι σχετικά σημαντική και γι' αυτό και η πολιτική συνοχή είναι πολύ σημαντική για τι μικρέ επιχειρήσει, αλλά και για όλε τι ε, ε, ενώσει, οργανώσει και διοικητικού μηχανισμού που στόχο έχουν να μειώσουν την ανεργία. Είναι λοιπόν δυνατόν να υπάρξει μια πολιτική που να δίνει την πρόσβαση στους πόρους. Αυτό δεν ε, θα είχε καταστεί δυνατό αν δεν είχαμε την ε, πρόσβαση στα διευθυντικά ταμεία. Δυστυχώς όμως τα αποτελέσματα, οι επιδόσεις μας, αν και είναι αξιοσημείωτα, δεν μπόρεσαν όλοι να ωφεληθούν ε, το ίδιο. Είναι σημαντική η στήριξη αυτή για μας και άκουσα και την ε, γερουσιαστή από την Λιθουανία. Η Σουηδία είναι μια από τις πιο βόρειες χώρες και για όντως για μας η Λιθουανία αποτελεί εξαιρετικό ε, ε, παράδειγμα όσον αφορά την απλοποίηση των διαδικασιών έτσι ώστε να μπορέσουν όσοι έχουν μικρά προγράμματα να έχουν και αυτή πρόσβαση στους πόρους. Πολύ θα ήθελα και εμείς να μπορέσουμε έτσι να απλοποιήσουμε τις διάφορες διαδικασίες ε, αυτοί οι οποίοι θα πρέπει να ασκήσουν αυτή την πολιτική είναι κυρίως οι επιχειρήσεις οι οποίες είναι εγκατεστημένες στις περιοχές μας. Εγώ έχω συναντήσει διάφορους ε, επιχειρηματίες που σήμερα ανησυχούν για τη δυσκολία αλλά και για την αβεβαιότητα όσον αφορά την πρόσβαση στα προγράμματα γιατί όπως μου λένε είναι δύσκολο κανείς να έχει πρόσβαση στα κονδύλια αυτά. Πρέπει να έχει πολύ μεγαλύτερο κεφάλαιο από αυτό ε, το οποίο έχει στη διάθεσή του και έπειτα δεν γνωρίζουν ακριβώς πώς πρέπει να συμπεριφερθούν. Και φυσικά όλα αυτά αποτελούν πρόβλημα για πολλοί κόσμο. Σίγουρα προσπαθήσαμε να χρησιμοποιήσουμε καλύτερα τα κονδύλια. Υπήρξαν μάλιστα και προγράμματα για τα οποία έγιναν ε, ε, για τα οποία υπήρξαν προβλήματα. Ε, πολλές φορές δηλαδή οι πληρωμές ήταν λιγότερες από αυτές που είχαν προβλεφθεί και ήταν πολύ δύσκολο για τους επιχειρηματίες να καλύψουν τη διαφορά χρηματοδότησης. Αυτό παρά το γεγονό ότι η διαφορά χρηματοδότηση ανάμεσα στην ίδια χρηματοδότηση και την κοινοτική δεν οφείλεται σε κάτι ε, παράνομο. Μιλάμε για προθεσμίες, για ε, προθεσμίες καταβολής των ποσών κτλ. Πολλές φορές είναι λίγα χρήματα. Πάντως είναι αυτός ο κόσμος ο οποίος στην ουσία θέτει σε εφαρμογή τις πολιτικές μας. Γιατί χωρίς αυτούς τους μικροεπιχειρηματίες όλα αυτά τα προγράμματα που θέλουμε να κάνουμε δεν θα υλοποιηθούν. Ελπίζω πως η Σουηδία λοιπόν θα μπορέσει να ασκήσει την αυτοκριτική της. Η Λιθουανία μας έδειξε τελευταία και το πώς θα πρέπει να προχωρήσουμε, πώς πρέπει να φερθούμε και ελπίζω πραγματικά πως η Σουηδία θα εκμεταλλευτεί αυτό το παράδειγμα, θα αποκομίσει διδάγματα και θα μπορέσει να τα καταφέρει καλύτερα, κυρίως για όσους πρέπει να εργαστούν σε αυτόν τον τομέα. Έχουμε πολλά να μάθουμε λοιπόν από τη Λιθουανία. Σας ευχαριστώ. Πρόεδρο, σας ευχαριστώ και εγώ. Και τελευταίος ο που είναι εγγεγραμμένος. Μένουμε μάλιστα στη Σουηδία, αλλά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ο Γκέραν Φέρμα. Ε, σας ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Δυστυχώς δεν μπόρεσα να είμαι παρόν καθ' όλη τη διάρκεια του εργαστηρίου λόγω άλλων δεσμεύσεων και υποχρεώσεων συνδέονται δε με αυτό με ε, το για το οποίο μίλησε ο Πολωνός συνάδελφος γιατί έχουμε το συναδέλφους της Euronest και τον πρόεδρο της Euronest σε μια πολύ σημαντική συνεδρία σήμερα εδώ που αφορά υποδομές και εμπορικές συμφωνίες με τους ανατολικούς μας γείτονες και αυτό έχει σχέση με τον ευρωπαϊκό προπολογισμό. Αναφέρομαι στην κυρία Νορδέρ που μίλησε πριν από μένα και είπε ότι υπήρξαν πολλές εντάσεις στις ε, συζητήσεις για τον προϋπολογισμό και αυτό είναι βέβαια αληθές. Όταν λοιπόν θα περάσουμε στο μέλλον από αυτή τη διαδικασία για το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο, το οποίο μόλις ολοκληρώσαμε, θα πρέπει να σκεφτούμε τι προκάλεσε αυτά τα προβλήματα. Πολλά από αυτά τα προβλήματα ήταν πιο πολύ πολιτική φύση και όχι οικονομική ή δημοσιονομική. Και αυτό ελπίζω στο μέλλον να το ξεπεράσουμε. Τώρα, όταν μιλάμε για την μέση ενδιάμεση αναθεώρηση αυτού του πολιετού ή του επόμενου θα πρέπει να σκεφτούμε πολλά πράγματα. Καταρχήν θα πρέπει να συμφωνήσουμε τα κράτη-μέλη και τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα ότι βασικό στο... έμφαση θα πρέπει να δοθεί στου τομεί όπου έχουμε ε, προστιθέμενη ευρωπαϊκή αξία. Γιατί εκεί θα πρέπει να είμαστε πιο φιλόδοξοι από ό,τι μέχρι τώρα, διότι οι προκλήσει είναι τεραστίων διαστάσεων θα πρέπει να δει κανεί τον παγκόσμιο ανταγωνισμό, έρευνα και ανάπτυξη. Αν θέλουμε να είμαστε πρωτοπόροι παγκοσμίω, κανένα ευρωπαϊκό κράτο δεν μπορεί να τα καταφέρει μόνο του. Πρέπει να συνεργαστούμε και να κάνουμε και πολύ περισσότερα από όσα κάνουμε μέχρι τώρα. Και αυτό πολιτικό δεν θα πρέπει να είναι επίμαχο ζήτημα. Δυστυχώ όμω φτάσαμε σε ένα δημοσιονομικό πλαίσιο που λέει ναι, υπάρχει αύξηση στην έρευνα και στην ανάπτυξη, αλλά μόνο μετά το 2016. Δηλαδή άλλα τρία χρόνια προπολογισμού σε αυτό το νέο δημοσιονομικό πλαίσιο χωρίς καμία αύξηση σε σχέση με το 2013 όσον αφορά την έρευνα και την ανάπτυξη και αυτό πραγματικά είναι πολιτική καταστροφή. Και μπορεί κανείς να δει και τι γίνεται με την πολιτική γυτνίασης. Έχουμε μια τεράστια πρόκληση προς, με τους γείτονες προς Νότο. Κοιτάξτε τη διάσκεψη που κάνουν τώρα στην Ελβετία για τη Συρία. Πιστεύει κανείς ότι θα ξεφύγουμε από αυτή την κατάσταση χωρίς ουσιαστική ευρωπαϊκή συμβολή για να οικοδομηθεί το μέλλον για χώρες όπως η Συρία ή η Προσανατολάς, άλλοι γείτονες. Αναφέρθηκε η Ουκρανία και η δύσκολη κατάσταση στη Μολδαβία ή αλλού. Πιστεύει κανείς πραγματικά πως θα βγούμε από αυτή την κατάσταση χωρίς μια ουσιαστική συμβολή από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την κατασκευή υποδομών, για την κατασκευή ενός οικονομικού μέλλοντος. Αν δεν το κάνουμε εμείς θα το κάνουν άλλοι. Και αυτό θα έχει πολιτικό αντίκτυπο. Είναι εξαιρετικά σημαντικό λοιπόν να σκεφτούμε τον προπολογισμό της Ένωσης Υπό αυτού του όρου. Από την άλλη πλευρά, βεβαίω, αυτό σημαίνει επίση πω αν δώσουμε πραγματικά προτεραιότητα σε όλα αυτά, υπάρχουν άλλα πράγματα τα οποία θα χάσουν την προτεραιότητά του. Και ίσω θα πρέπει να είμαστε λίγο αυτοκριτικοί και να διερωτηθούμε αν υπάρχουν τομεί που μπορούν να περικοπούν ή να είναι πιο αποτελεσματική η δράση μα εκεί. Αλλά πιστεύω πραγματικά πω τα κρατή-μέλη θα πρέπει να εξετάσουν το θέμα τη χρήση του προπολογισμού τη Ένωση ω ένα μέσο για να βρουν εξοικονομία μίση μάλλον για τι ίδιε. Α δούμε την υπηρεσία εξωτερική για παράδειγμα. Και εγώ ήμουν ένα από του ηγητέ στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων για την Υπηρεσία εξωτερική δράση. Η ιδέα είναι πω η νέα αυτή υπηρεσία θα πρέπει να καταστήσει δυνατή την αποταμίευση, την εξοικονόμηση για τι εθνικέ υπηρεσίε εξωτερικών υποθέσεων. Αλλά έχω την εντύπωση ότι Πάει ανάποδα το πράγμα. Ότι χρειάζονται και προσλαμβάνουν περισσότερο κόσμο στα Υπουργεία Εξωτερικών για να παρακολουθεί τι συμβαίνει στι Βρυξέλλες. Νομίζω λοιπόν πως πρέπει να, να αναζητήσουμε τις δυνατότητες για εξοικονομήσεις στον ευρωπαϊκό προπολογισμό. Ας δούμε λοιπόν τι θα μπορέσουμε να κάνουμε ε, με αυτές τις εμπειρίες από αυτή τη διαδικασία και να τη βελτιώσουμε για το μέλλον. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ Γκέραν. Θα ζητήσω τώρα από τους συναδέλφους εδώ, αν θέλουν τον λόγο, ιδίως ε, προς την Κομισιόν στην οποία τέθηκαν πολλές ερωτήσεις. Θέλω να ρωτήσω τα μέλη του Προεδρείου αν θέλουν να μιλήσουν πρώτα η Κομισιόν. Ευχαριστώ. Να ευχαριστήσω τους άλλους συναδέλφους που έκαναν παρουσιάσεις και όλους όσους μίλησαν για... αναγνώρισε ότι η πολιτική συνοχή διαδραματεί σημαντικό ρόλο για την ανάπτυξη και την ε, απασχόληση και τα παραδείγματα που αναφέρατε με χαροποιούν ιδιαίτερως. Αλλά ευχαριστώ και για τα πιο κριτικά σχόλια. Κάτι που αποδεικνύει ότι φυσικά υπάρχει περιθώριο για βελτιώσεις. Πολλοί ομιλητέ αναφέρθηκαν στην ανάγκη απλούστευσης. Και είναι αλήθεια ότι οι κανόνες είναι περίπλοκοι. Και είναι σημαντικό τουλάχιστον αν έχουμε περίπλοκους κανόνες, να έχουμε μόνο μία δέσμη κανόνων. Και αυτό καταφέραμε για την επόμενη περίοδο, να έχουμε πέντε μεν μία, αλλά ένα πλέγμα κανόνων, μία δέσμη κανόνων. Αυτό από μόνο του διευκολύνει τα πράγματα. Θα πρέπει επίσης ε, να έχουμε κατά νου ότι θα πρέπει να φροντίσουμε να είναι σωστή η αξιοποίηση των κονδυλίων, να είναι τακτική, κανονική, χωρίς ατασταλίες και να γίνεται και ο έλεγχος. Και αν υπάρχουν αποδείξεις ότι κάποιος δεν τήρησε τους κανόνες κρατικών προμηθειών, θα πρέπει να γίνει μία διόρθωση οικονομική. Θα πρέπει να φροντίσουμε ώστε τα κονδύλια να αξιοποιούνται για το σκοπό που προβλέφθηκαν και φυσικά με τήρηση των κανόνων. Στην αρχή είχαμε μία παρέμβαση για την εκτέλεση. Ο κύριος Γκοτσμάνης έχει φύγει στο μεταξύ, αλλά δεν θα ήθελα να αφήσω αναπάντητα τα σχόλιά του. Καταρχήν τα ραλ, τα ρέστε τα υπόλοιπα προς εκαθάριση και μελλοντικές πληρωμές. Σε μία, έχουμε, σε μια πολιτική που είναι παιδιτική πολιτική, τα ράλ είναι κάτι το φυσιολογικό. Ακριβώς επειδή μιλούμε για επενδύσεις, ε, δεν, γίνεται, δεν συγκεντρώνονται όλες οι πληρωμές σε μία χρονιά, μετακυλίονται για την επόμενη. Γι' αυτό και έχουμε ραλ. Υπόλοιπα προς εκαθάριση. Βέβαια δεν θέλουμε υπερβολικό αριθμό ραλ. Κάτι τέτοιο είναι ανεπιθύμητο. Και στην πολιτική μας ακριβώς προβλέψαμε κάποιους περιορισμούς για να περιχαρακώσουμε τα ραλ. Έχουμε τον νη ε, συν 2 και το περίφημο νη συν 3. Αρχικά είχαμε προτείνει νη συν 2 στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τώρα έχουμε νη συν 3, κάτι που αύξησε τα ράλ. Στις εισαγωγικέ μου παρατηρήσεις έκανα ε, μια ανοίξη για το πρόβλημα αυτό και την πίεση στις πληρωμές. Και δεν είναι μυστικό ότι η εκτέλεση ποικίλει από χώρα σε χώρα. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι πέρασε απαρατήρητο το θέμα από μας ότι το παραβλέψαμε. Και η βασική αιτία της χαμηλής εκταμίευσης, της χαμηλής απορρόφησης, είναι η ελληπής δημοσιο... ικανότητα του δημοσίου στα διάφορα στάδια της εφαρμογής. Από τη χάραξη των τομεακών πολιτικών, υδροδότησης, μεταφορών. Μερικές φορές δεν υπάρχει εκεί διοικητική ικανότητα για την ε, χάραξη, σχεδιασμό των προγραμμάτων, ε, επιλογή των προγραμμάτων, οργάνωση διαγωνισμού για τις κρατικές προμήθειες και ούτω καθεξής. Αναγνωρίσαμε αυτές τις ε, δυσκολίες και ως Γενικός Διευθυντής, ακόμη και με μειωμένο προσωπικό, αυτά που προσπαθήσαμε στην τελευταία διοργάνωση να δημιουργήσουμε μια νέα μονάδα που ασχολείται ακριβώς με την ενίσχυση των διοικητικών θεσμών, ώστε χώρες που υστερούν στην εκταμίευση να καλύψουν το χαμένο έδαφος, να ενισχύσουν τις διοικητικές τους δομές. Ζητήσαμε και τη στήριξη της Παγκόσμιας Τράπεζας και άλλων διεθνών οργανώσεων για να βοηθήσουμε στη χάραξη των μεακών στρατηγικών. Δεν είναι λοιπόν ότι δεν αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα και στην επόμενη περίοδο προγραμματισμού θα επικεντρωθούμε ιδιαίτερα στα θέματα αυτά και στο ζήτημα της καταπολέμησης της διαφθοράς και δωροδοκίας. Αναφέρθηκε προς ανατολισμό στα αποτελέσματα και η ανάγκη θέσπισης κάποιων δικτών. Συμφωνώ απολύτως. Αυτή τη στιγμή έχουμε απορροφηθεί από τη λογική της εκταμίευσης. Μας ενδιαφέρει πόσα κονδύλια εκταμιεύθηκαν και ποιο είναι το ποσοστό απορρόφηση, αλλά μας ενδιαφέρει επίσης αν υλοποιήθηκαν οι στόχοι. Και στο μέλλον θα έχουμε νομικό πλαίσιο που θα υποχρεώνει τα κράτη-μέλη και τις περιφέρειες να ενημερώνουν τακτικά για τα επιτεύγματά τους, για το βαθμό υλοποίηση των στόχων. Και μάλιστα όλα αυτά τα στοιχεία θα είναι δημόσια, ώστε ο καθένας θα μπορεί να ελέγξει όχι μόνο πόσα κονδύλια εκταμιεύθηκαν, αλλά και τι επιτεύχθηκε στην πράξη. Το θέμα της μακροαιρεσιμότητας. Θα μπορούσαμε να έχουμε ένα ολόκληρο σεμινάριο μόνο για αυτό το θέμα. Πάντως, ε, είμαι πεπισμένος ότι εφόσον η πολιτική συνοχή θέλει να διαδραματίσει ρόλο το σύνολο της οικονομικής πολιτικής και να συνεχίσει να έχει σημαντικό προϋπολογισμό θα πρέπει και η πολιτική συνοχής να στηρίζει, να σέβεται την διασύνδεση που υπάρχει μεταξύ των τριών κορυφών του τριγώνου. Γιατί αν δεν είναι υγιεί τα δημόσια οικονομικά, δεν θα δημιουργούνται, δεν θα δημιουργούνται πρόσφορες συνθήκες για την ανάπτυξη. Αν έχουμε υψηλά επιτόκια θα δημιουργούνται προβλήματα για οικονομικά για τις επιχειρήσεις. Όλα αυτά τα θέματα είναι αλληλένδετα. Αυτός ο σύνδεσμος, η διασύνδεση θα πρέπει να αναγνωριστεί και γι' αυτό και οι σχετικές διατάξεις θα πρέπει να λαμβάνουν αυτή τη διασύνδεση υπόψη. Τώρα, η αποσύνδεση της ανάπτυξης από το θέμα του στόχου διοξιδίου του άνθρακα. Αν ε, μελετήσετε τις προτεραιότητες που σας ανέφερα, θα λέγατε ότι, μια, η οικονομία με χαμηλές εκπομπές άνθρακα είναι από τις βασικές μας προτεραιότητες. Και εκεί θέλουμε να επικεντρώσουμε τα κονδύλια ανάλογα με την ε, κατηγορία στην οποία ανήκει η περιφέρειά σας. Τώρα, αν εξετάσουμε πιο εξονυχιστικά το μηχανισμό συγκέντρωσης, διαπιστώνουμε ότι υπάρχουν ειδικέ διατάξεις για τη μείωση διοξιδίου του άνθρακα. Οπότε υπάρχει σαφής πρόβλεψη στο νέο πλαίσιο. Είναι σαφές ότι η ενεργειακή αποδοτικότητα και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι σημαντικός κινητήριος μοχλός της ανάπτυξης αλλά και της προστασίας του περιβάλλοντος. Κύριε Πρόεδρε, αυτά και πιστεύω ότι απάντησα στις ερωτήσεις που μου τέθηκαν. Ευχαριστώ. Θέλετε κι εσείς να προσθέσετε κάτι? Um, Οι συνάδελφοι από την Πολωνία αναφέρθηκαν στην Ουκρανία. και ένας συνάδελφος ε, μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Δεν είναι δυνατόν να προχωρήσει η Ανατολική Γειτονία χωρίς στήριξη από τον ε, ενωσιακό προϋπολογισμό. Πρέπει να συνεχιστεί αυτή η προσπάθεια, Διαπραγματεύσει με την Ουκρανία, στήριξη για την Γεωργία. Γιατί αν θέλουμε μια δημοκρατική Ευρώπη πρέπει να στηρίξουμε αυτή την προσπάθεια. Συμφωνώ με τους συναδέλφους που αναφέρθηκαν στην ανάγκη απλούστευσης των κανόνων και διαδικασιών και την ε, μείωση της γραφειοκρατίας. και από πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Γιατί ξέρετε, σε κάποιες περιπτώσεις διάφοροι εμπειρογνώμονες εγκαταλείπουν την προσπάθεια αξιοποίησης των ε, διαθροτικών ταμείων γιατί είναι πολύ περίπλοκο, παίρνει πολύ χρόνο και ξέρετε η επιστήμη ε, εξελίσσεται πολύ πιο γρήγορα από τις διαδικασίες και οι κανόνες για τις δημόσιες προμήθειες. Όλα αυτά ε, πολλές φορές οδηγούν στο να πληρώνουν ε, οι, δήμοι μας τα σπασμένα διότι έχουν μεγάλο χρέος. Ιδίω περιβαλλοντικά προβλήματα. Τώρα, ποιοι θα είναι οι στρατηγικοί προσανατολισμοί για την επόμενη περίοδο. Η αναβιομηχάνηση της Ευρώπης είναι το κύριο, αν θέλουμε περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας. Το βασικό πρόβλημα για την αναβιομηχάνηση είναι ότι οι νέες βιομηχανίες πρέπει να βασίζονται στην έρευνα και την καινοτομία. Αυτή θα, θα πρέπει να είναι η βασική μας κατεύθυνση και η ενεργειακή αποδοτικότητα, βεβαίως. Σε σύγκριση με τις Ηνωμένε Πολιτείες, υπολοιπόμεθα. Διότι οι ενεργειακοί πόροι των ΗΠΑ ε, είναι στο 50% ε, της τιμής των δικών μας. Άρα αυτό θίγει την ανταγωνιστικότητά μας. Η αποτελεσματικότητα και η αποδοτικότητα της ενεργειακής χρήσης πρέπει να είναι βασική προτεραιότητα για την επόμενη περίοδο. Και... Όχι. Και τίποτα άλλο. Αυτά ήθελα να πω. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρος. Η Μαρία. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δύο λεπτάκια για να αναπτύξω μια ιδέα που θεωρώ θεμελιώδη και άλλωστε την ανέφεραν και πολλοί προλαλήσαντες. Ε, πρόκειται για τη σωστή αξιοποίηση των πόρων. Μας είπε ο Γενικός Διευθυντής ε, ότι χωρίς υγιή δημόσια οικονομικά δεν νοείται ανάπτυξη. Και θα ήθελα να επιμείνω σε αυτό και να αποτίσω φόρο τιμή στις τεράστιες προσπάθειες που κάνουν ορισμένε χώρες και ιδιαίτερα τις προσπάθειες της Ισπανίας για δημοσιονομική εξυγίαση, για σταθεροποίηση των δημόσιων οικονομικών και για τη συμμόρφωση με τις ανηλυμένες υποχρεώσεις. Χάρη σε αυτή την προσπάθεια καταφέραμε σε μεγάλο βαθμό να έχουμε τα αποτελέσματα που ανέφερε ο πρόσωπος Ευρωπαϊκής Επιτροπή. Και σας ευχαριστώ, μας είπε για την ε, θαραλέα απόφαση της Ισπανικής κυβέρνησης. Και η σωστή αξιοποίηση των πόρων εξαρτάται από τη σωστή εξασφάλιση των προϋποθέσεων. Θα πρέπει να γίνουν οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις ε, προηγουμένως. Στην Ισπανία έχουμε επιφέρει περίπου 100 μεταρρυθμίσεις. Νομίζω ότι κάνουμε ό,τι μπορούμε για να εφαρμόσουμε όχι μόνο τη δημοσιονομική εξυγίανση, και να εξασφαλίσουμε τη βιωσιμότητα των συντάξεων, όχι μόνο να μεταρρυθμίσουμε την εκπαίδευση και να, να καταπολεμήσουμε την ε, εγκατάλειψη της φίτησης, αλλά θέλουμε και βραχυπρόθεσμες μεταρρυθμίσεις, προκειμένου να δώσουμε νέα πνοή και σημαντικά ενάψματα στις επενδύσεις, στο επιχειρηματικό πνεύμα και στην ε, εφαρμογή νέων πρωτοβουλειών και ανασυγκρότηση του παραγωγικού ιστού. Γιατί όπως σας είπα έκλεισαν περίπου μισό εκατομμύριο επιχειρήσεις μεταξύ 2008 και 2011. Θα πρέπει αυτόν τον ιστό να τον αποκαταστήσουμε, να τον επουλώσουμε. Επίσης η σωστή αξιοποίηση των, φόρων, των πόρων συγγνώμη, σχετίζεται με την ευελιξία, την προσαρμοστικότητα και τον προγραμματισμό και επαναπροσανατολισμό των κονδύλιων αυτών. Όλα αυτά τα στοιχεία τα αξιοποίησαμε στην Ισπανία και επικεντρωθήκαμε στις βασικότερες προτεραιότητες ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες και τις διαρθρωτικές αδυναμίες της πατρίδας μου. Γιατί μίσον στόχος ήταν η καταπολέμηση της ανεργίας και κυρίως της ανεργίας των νέων. Επίσης, θέλησαμε να αποκαταστήσουμε την ροή της χρηματοδότησης προς τους αυτοαποσχολούμενους και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Είναι απαραίτητο και στο μέλλον να διασφαλίσουμε και να διατηρήσουμε αυτή την προσαρμοστικότητα και την ευελιξία των διαρθρωτικών κονδυλίων στις ε, ανάγκες και στα προβλήματα. Φυσικά εφαρμόζοντας και εμείς τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις ε, σε συνεργασία όμως με την πολιτική συνοχής. Έτσι θα επενδύσουμε ουσιαστικά στο μέλλον ώστε να αντιληφθούν και οι συμπολίτες μας ότι και η Ευρώπη είναι ευαίσθητα στα προβλήματά τους και επιλύει καθημερινά όλο και περισσότερα. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, θέλετε να αντλήσετε τα συμπεράσματα από την πρωινή συζήτηση. Θέλω να σας ευχαριστήσω για την συνεργασία της συνδιοργάνωσης της σημερινής εκδήλωσης. Ε, θέλω να ευχαριστήσω τους ομιλητές του πάνελ αλλά και όλους τους εκπροσώπους των Εθνικών Κοινοβουλίων ή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που πήραν το λόγο και κατέθεσαν τις απόψεις τους για το μέλλον των πολιτικών συνοχής. Η μεγαλύτερη πρόκληση για την Ευρωπαϊκή Ένωση στα ερχόμενα χρόνια είναι να διασφαλίσει συνθήκες βιώσιμης ανάπτυξης στις χώρες μέλη, προϋπόθεση για δημιουργία θέσεων εργασίας. Αυτός είναι ο μόνος ασφαλής τρόπος για την καταπολέμηση της ανεργίας και την διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής. Η αύξηση της ανεργίας και η ενίσχυση των κοινωνικών ανισοτήτων δημιουργούν απειλές για το πολιτικό μας σύστημα και ενισχύουν τον ευρωσκεπτικισμό. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η άνοδος των νεοναζιστών στην Ελλάδα. Η αντιμετώπιση της κρίσης προϋποθέτει πόρους, αλλά δεν έχουμε τόσους όσους χρειαζόμαστε. Άρα θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί στην αξιοποίηση αυτών των πόρων που έχουμε θα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι οι κοινοτικοί πόροι συνοχής συμβάλλουν όχι μόνο στην ανάπτυξη, αλλά βοηθούν και στη μείωση των ανισοτήτων μεταξύ των περιφερειών αλλά και μεταξύ των χωρών. Επισημένω αυτό που είπε και ο κύριος Ντεεφά, παρά τους πόρους που διατέθηκαν, δεν καταφέραμε να μειώσουμε τις ανισότητες μεταξύ των περιφερειών. Αυτή θα είναι η μεγάλη πρόκληση για τη νέα προγραμματική περίοδο. Και εδώ η περαιτέρω συνεργασία Εθνικών Κοινοβουλίων και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μπορεί να βοηθήσει καθοριστικά. Αυτή είναι η θέση του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Προς αυτή την κατεύθυνση θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε και οι διακοινοβουλευτικές διασκέψεις όπως η σημερινή βοηθούν προς αυτή την κατεύθυνση. Σας ευχαριστώ πολύ. Πολύ ωραία. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα λοιπόν να νέου ευχαριστήσω τον Πρόεδρο, τα μέλη του, των, της ομάδας των ομιλητών και όσους συμμετείχαν σε αυτή την ανταλλαγή απόψεων είδαμε ποια ήταν τα κοινά σημεία, οι ελπίδες που μπορούμε να έχουμε από το νέο πλαίσιο, το νέο καθεστώς, διαπιστώνοντας πως δυστυχώς κάποια από τα προβλήματα θα παραμείνουν παρά τις προσπάθειες απλοποίησης. Βλέπουμε πως και αυτές οι προσπάθειες έχουν τα ωριά τους. Αυτό μας το έδειξε κυρίως η ε, ανταλλαγή ανάμεσα στους εκπροσώπους της ε, Λιθουανίας και της Σουηδίας. Μπορούμε να εμπνευστούμε από τις καλές πρακτικές ορισμένων χωρών και να τις χρησιμοποιήσουμε σε άλλες χώρες. Ε, το πρώτο πλονέκτημα το οποίο αποκομίζουμε από το γεγονός ότι συμμετέχουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι το να συζούμε σαν μέλη μιας οικογένειας και να μπορούμε να συγκρίνουμε τι πετυχαίνει, τι πάει καλά για τον ένα για τον άλλον. Όλος παραδόξως δεν είναι αυτό η πρώτη μας αντίδραση, το πρώτο μας αντανακλαστικό. Στην Ευρωπαϊκή συζήτηση συχνά έχουμε πολιτική συζήτηση για να δούμε αν χρειάζεται περισσότερη Ευρώπη ή λιγότερη Ευρώπη. Είναι μια σημαντική συζήτηση αυτή. Ωστόσο δεν αφιερώνουμε αρκετά το προβληματισμό μας στο θέμα του πώς καλύτερα θα εκμεταλλευτούμε το γεγονός ότι συμβιώνουμε και στον τομέα που βασικά εμπίπτει σε την εθνική ευθύνη, δηλαδή φορολογία, ε, εθνική οικονομία κτλ. Θα πρέπει να κάνουμε καλύτερα τα όσα εξαρτώνται από την Ένωση, αλλά και να προσπαθήσουμε να εμπνευστούμε από αυτά που πέτυχαν στη γειτονική μας χώρα και πιστεύω πως τέτοιου είδους διασκέψεις συμβάλλουν σε αυτά όλα. Ευχαριστώ λοιπόν όλους τους ε, συμμετέχοντες και εδώ προτείνω να διακόψουμε τις εργασίες μας, να σταματήσουμε αυτή το εργαστήριο και να τα ξαναπούμε σε 10 λεπτά στην αίθουσα της Ολομέλειας που είναι στο τρίτο όροφο, αλλά από την άλλη πλευρά, στο άλλο κτίριο που ήμασταν χτέ και τη Δευτέρα, για να α, τα τελικά συμπεράσματα του συνόλου της διάσκεψης. Πέρα της συνεδρίαση.